Good morning. Καλημέρα σας, λέει ο πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Good to see you all back to work to be back. Χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε μετά τις διακοπές και ελπίζω ότι περάσατε όλοι καλά. Και ξεκινούμε μια γεμάτη θέματα ημέρα στη διάταξη με την έγκρισή της. έχετε λάβει θα πρέπει να προσθεθεί ένα σημείο η έγκριση του προσθετικού κατόπιν ε, της δουλειάς που έκαναν οι Ρωσομαθισμομικοί όσον αφορά το Σέγγεν για την έκθεση κυρίας Μπέβα. Όπως το, και θα το συζητήσουμε αργότερα. Υπάρχει κάποια ένσταση. Επομένως θεωρώ ότι την εγκρίνεται πάνω στο σημείο παριθμών 2, δηλαδή έγκριση των συστάσεων των συντονιστών που έχουν ως εξής πρώτα-πρώτα τον ορισμό εισηγητών, η κυρία Φαζόν, όσον αφορά το, το προστατευμένο καθεστώ για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, εκείνη επί τη βάση της μονομέρους αναγνώριση από Κροατία, Κύπρο κάποιων εγγράφων. Αναφέρονται εδώ πέρα κατά λεπτό και κατόπιν έχουμε την έκθεση του κυρίου Μωράε. Είναι ο εισηγητή για το πρόγραμμα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΗΠΑ. Εγκρίνονται οι προτάσεις των εισηγητών και στη συνέχεια έχουμε το διορθωτικό. Το... Τη δέσμη μέτρων διακυβέρνηση του Σέγγεν θα ακολουθεί τη ε, Βέμπερ και σύμφωνα με τι διατάξει του κανονισμού 216 αυτά πρόκειται να ζητούν μετά την ψήφιση στην Ολομέλεια. Οι μεταβολέ εδώ είναι κλασικά, αποκλειστικά γλωσσικού χαρακτήρα, δεν έχετε ενστάσει. Θεωρούμε ότι το διορθωτικό εγκρίνεται. The, uh, mention on the delegation to Greece. Έχουμε την έκθεση την απολογιστική που αφορά την ε, αντιπροσωπεία μας στην Ελλάδα του Ιουλίου και ε, αυτό το κείμενο θεωρούμε ότι εγκρίνεται κατόπιν έχουμε τώρα την έγκριση των πρακτικών Οκτωβρίου, Ιανουαρίου του 2013. Τρεις συνδυάσεις. Και αν μέχρι το πέρας της συνδυάσεις δεν έχουμε ενστάσεις, τότε θεωρούμε ότι αυτά τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Και τώρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και σας υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να έχετε τις ε, κάρτες της ψηφοφορίας για να κάνουμε τον ε, έλεγχο όποτε χρειάζεται. ψηφίσουν αυτοί που δικαιούνται να ψηφίσουν και αν δεν έχετε αντίρρηση προχωρούμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το γενικό προπολογισμό του 2014 ε, όλα τα τμήματα αυτού. Πρώτα πρώτα θα ψηφίσουμε. Τζαν Μούλτερ, Τζαν Μούλτερ, Έκθεση Mulder. Έκθεση Μίλτερ που αφορά την κρίση 2014. Αφορά το σχέδιο προπολογισμού και προχωρούμε επομένω στην ψηφοφορία. Okay. I am going to announce the amendments as usual. Θα σας λέω ποιες τροπολογίες ψηφίζουμε, ως συνήθως. Amendment 61-0-0. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 61-0-1. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 61-02, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 6103 υπέρ κατά απορρίπτεται 6104 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος ε, ο πρώτης όποιος εγκρίνεται αλλά θα ελέγξουμε έλεγχος ψηφίζουμε τώρα

κατά, απορρίπτεται, 1.07. υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 6108, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται, Έχουμε μια προφορική τροπότητα τελευταία στιγμή και είπαμε ότι εδώ έχουμε ζητήσει για τη ΣΕΜΠΟΛ ένα νέο ποσό 8 εκατομμύρια 450.640. Δηλαδή ε, ε, φτάσουμε στο επίπεδο της επίσης υποχρεώσεων του 2013. Υπάρχει κάποια ένσταση. Ψηφίζουμε το 6109. Υπέρ. Κατά. 61, 6110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6111. Υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61-14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61-15 υπέρ κατά αποχές πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος Ξανά 15 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφοφορίας. 20-25 απορρίπτεται. 61-16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-17 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος, εκ πρώτης όψης απορρίπτεται, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, πέρας, 21-25, Εξτένα 61-17, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος 61-19, κατά, αποχέ, απορρίπτεται, 61, 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61, 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61, 21. Ταυτόσημη. Ξεντένα 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Λειτουργικός έλεγχος του 61-23. Πέρας. Και απορρίπτεται. 61-24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει έλεγχος. 20, για την 61, 24. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. 25, 21 εγκρίνεται. Five. Favor. 61-25 υπέρ κατά αποχές και απορρίπτεται 61-26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στένα 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, όχι. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Συμπαθάτε με. Στένα 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61-31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε έλεγχο στην 61-31. Ψήφιζουν. Πέρας. 23-25 απορρίπτεται. 61-32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ξένα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. Και γίνει ηλεκτρονικό έλεγχο. Το 61-33. Ψηφίζουμε. Ναι, απορρίπτωτα. 22, 26. Και τώρα. 61, 34. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Και 35. υπέρ Απορρίπτωτα. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότηση του κυρίου Μούλτερ. Πρώτο απολογία. Υπέρ. Κατά. Απογές. Εγκρίνεται. Δεύτερη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Έλεγχος. Και κάνω λιτρό έλεγχο για την τροπολογία δύο. Ψηφίζουμε. No, I'm sorry, it was rejected. 23. 23-26 απορρίφθηκε. Τρίτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές οριακό το αποτέλεσμα αποφύγουμε τα λάθη, να κάνουμε έλεγχο. Τέσσερα ψηφίζουμε. Τι έχουμε. Πέρασε. 17.31. Σαφώς απολύπτεται. Και τώρα. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά.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 Ψηφίζουμε. Πέρας. 24-25. Άρα απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, ψηφίζουμε τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Μίλτος. Α, μάλιστα λέω πρόεδρος. Έγινε η ψηφοφορία. I really Thank you, thank you all. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Παρακαλώ όσοι ήταν να το κάνετε γρήγορα. Do it gently so that we can move on to the following point. Let let Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα, αλλά να μου επιτρέψετε πρώτα να αναφερθώ για την κατάσταση των εξελίξεων, των διαπραγματεύσεων και των νομοθετικών διαδικασιών. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Aquí eh, Λοιπόν, να επανέρχομαι στο που βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και των νομοθετικών διαδικασιών. Για το θέμα Μακοβέη, ο τριμερής διάλογος ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή χθες. Η κυρία Μακοβέη δεν είναι στην πόλη μας σήμερα και θα μας παρουσιάσει την κατάσταση των διαπραγματεύσεών της στην Επιτροπή μας στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της τακτικής μας συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στην κοινή συζήτηση σχετικά με τα σημεία 6 και 7. Το σημείο 6 είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρακαλώ λίγη σιωπή θα βοηθήσει. Περνάω, επαναλαμβάνω, λέει ο Πρόεδρος, στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με τα βήματα προόδου για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για τους Ρωμά. Και έχουμε στο σημείο 7 και τη σύσταση του Συμβουλίου για τα μέτρα ένταξης των Ρώμα στα κράτη-μέλη θα ακούσουμε την παρουσίαση την οποία θα μας κάνει ο Αβρίλιο Τσομπάνου Ντορντέα, Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ακολουθήσει ε, ανταλλαγή απόψεων. Η Επιτροπή εξέδωσε ένα ανακοινοθένος της το 2011 για τις στρατηγικές της εθνικές ένταξης των Ρωμά και ζήτησε από τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική σχετικά με ε, τις πολιτικές τους αυτές. Έχει εν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογήσει τις στρατηγικές αυτές, έχει κάνει συστάσεις και μετά από ένα χρόνο έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα ανακοίνωση για τα βήματα που έγιναν στα πλαίσια της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση του κυρίου Τζομπάνου Ντορντεά και μετά έχετε το λόγο εφόσον το επιθυμείτε. Κύριε Τζομπάνου Ντορντεά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δώσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τα έγγραφα τα οποία έγιναν σαν πακέτο δεκτά από το σύνολο των Επιτρόπων στο τέλος του Ιουνίου πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Όπως ξέρετε ότι το θέμα της ένταξης των Ρωμά είναι ε, σημαντική προτεραιότητα πολιτική της Επιτροπής και χάρη ακριβώς την αιμονή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Στο παρελθόν είχαν γίνει συζητήσεις και σε επίπεδο του Συμβουλίου και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε τον μήνα Ιούνιο νομίζω αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία για την συγκεκριμένη και συνεκτική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την συνεχή προσοχή την οποία δίδει η Επιτροπή στις προσπάθειες των κρατών μελών για την προώθηση της ένταξης των Ρωμά. Το πρώτο συνθετικό αν θέλετε του πακέτου της 26ης Ιουνίου είναι η ανακοίνωση η οποία στην ουσία είναι μια έκθεση αξιολόγησης ενός συνόλου διαφθρωτικών στοιχείων των πολιτικών των κρατών μελών. Ενθυμίστε ότι ήδη το 2012, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει μία σειρά διαφορετικών στοιχείων απαραίτητων για τη σωστή εφαρμογή των πολιτικών αυτών στρατηγικών. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ε, κατάλληλη χρηματοδότηση, ανάπτυξη παρακολούθησης των εφαρμοσμένων πολιτικών, ε, αυτό θα επιτρέψει και τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, ε, θα επιτρέψει την κατάργηση των διακρίσεων και θα δημιουργήσει και εθνικά σημεία συντονισμού των πολιτικών ένταξης των Ρωμά. Πέραν αυτών έχουμε και τα διαρθρωτικά μέτρα γιατί θεωρούμε ότι μια πραγματική πρόοδος στην ένταξη των Ρωμά στον τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας και της κατοικίας δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της, ε, ε, θα έλεγα, ε, του εφικτού χαρακτήρα αυτών των πολιτικών. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν εμείς να αναλαμβάνουμε τη μία μέρα μια υποχρέωση και να μην μπορούμε να την υπηρετήσουμε. Απαιτούνται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της πορείας της προόδου για τα επόμενα χρόνια. Αφιερώσαμε λοιπόν την έκθεση αξιολόγησης του μηνός Ιουνίου στην ανάλυση των δημάτων προόδου που έκαναν τα κράτη-μέλη ή που θα έπρεπε να είχαν κάνει μέσω της εφαρμογής των διαφθορτικών πολιτικών. Η αξιολόγησή μας δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ θετική. Ναι μεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος από ορισμένα κράτη-μέλη ε, τον προηγούμενο χρόνο μετά από τις συστάσεις τις οποίες κάναμε αλλά δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά επί τόπου. Κάθε κράτος μέλος έχει δημιουργήσει αυτό το εθνικό συντονιστικό αν ε, χώρο ο οποίος φροντίζει τα, της ένταξης των ε, Ρωμά και των πολιτικών αυτών Πολλές φορές όμως ε, αυτά τα κέντρα τα εθνικά δεν έχουν τα μέσα, τους πόρους και κυρίως δεν έχουν την πολιτική στήριξη που απαιτείται για την επίτευξη των καθηκόντων τους και των στόχων τους. Είναι επίσης αληθές ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πάρει μέτρα για να εμπλέξουν τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές ε, και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια του καθορισμού των μέτρων ένταξης των Ρωμά. Όμως παρατηρήσαμε ότι σπάνια η εμπλοκή αυτή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών παίρνει συστηματικό χαρακτήρα πάρα πολύ σπάνια και δεν βοηθά ε, την πολιτικές ε, ένταξης των Ρωμά. Η κατανομή των βασικών απαιτούμενων θα έλεγα οικονομικών πόρων είναι το πιο δύσκολο πράγμα για τα κράτη-μέλη, τα περισσότερα αν όχι όλα. Όταν αναφερόμαστε σε οικονομικούς πόρους ε, αναφερόμαστε κυρίως σε δημόσιες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό σε εθνικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αναφερόμαστε όμως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πιστώσεις που στοχεύουν στην ένταξη των Ρωμά, στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στις χώρες που αντιμετωπίζουν τα πιο σημαντικά προβλήματα στην ένταξη των Ρωμά. Πολλά έγιναν λοιπόν για την δημιουργία λειτουργικών συστημάτων παρακολούθησης της κατάστασης. Να, να παρατηρήσω εδώ ότι η υπηρεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει μια ομάδα παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών ένταξης Ρωμά. Συμμετέχουμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη σε εθελοντική βάση. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευρά των κρατών μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την ομάδα η οποία παρέχει ε, συμβουλευτική στήριξη αλλά στην ουσία η εφαρμογή των προτινομένων μέτρων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο των συστημάτων παρακολούθησης της κατάστασης δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Να μου επιτρέψετε λοιπόν εδώ να υπογραμμίσω ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό σημείο δυσκολίας, παρόμοιας δυσκολίας αν θέλετε με την ανάγκη κάλυψης των αναγκών με τους κατάλληλους πόρους. Η συνεχείς διακρίσεις και ο ρατσισμός που υφίστανται οι Ρωμά και η ανάγκη πραγματικής ουσιαστικής καταπολέμησης αυτών των εκδηλώσεων που εμφανίζονται σε πολλές χώρες. Οι διακρίσεις των Ρωμά στην παιδεία είναι διαδεδομένες σε πολλές χώρες. Όλες σχεδόν οι χώρες προωθούν, να, προωθούν την ένταξη των Ρωμά, αλλά αυτό απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα κάλυψης των αναγκών των μεμονωμένων πολιτών Ρωμά και απαιτεί συστηματικές παρεμβάσεις από πλευράς του νόμου και των αρχών καταστολής όταν αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε να διακοπούν συμπεριφορές απειλητικές, ρατσιστικές εις βάρος των πολιτών Ρωμά που είναι ε, ειρηνικοί και υπεύθυνοι πολίτες. Μετά από αυτή την σύντομη παρουσίαση λοιπόν των βασικών συμπερασμάτων της εκθέσεως που έγινε δεκτή τον μήνα Ιούνιο, να πω ότι στις αρχές του Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της μόνιμης ανησυχίας της για την σωστή εφαρμογή των μέτρων ένταξης έκανε ορισμένες συστάσεις αναχώρα τις οποίες πρότεινε στο Συμβούλιο και τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο στην καλοκαιρινή του συνάντηση στα πλαίσια της, Ευρώπης, ε, της διαδικασίας για την Ευρώπη 2020. Ε, Κάποιες συστάσεις αναχώρα λοιπόν αφορούν κυρίως πέντε χώρες θα έλεγα όπου η διάσταση της κοινότητας Ρωμά είναι μεγάλη και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές για την ένταξη των μελών της κοινότητας αυτής είναι, είναι πολύ σημαντικές. Αυτές οι συστάσεις αφορούν Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία. Uh, uh, Θα έπρεπε λοιπόν οι συστάσεις αυτές που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα και χώρες να είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιτικού πακέτου και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα περαιτέρω μέσο για να παρακολουθήσει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές τα κράτη-μέλη. Αυτή η ένταξη των ειδικών μέτρων στα πλαίσια του γενικότερου πακέτου έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι όπως γνωρίζετε οι πολιτικοί στόχοι οι οποίοι καθορίζονται από τις ε, ε, συστάσεις αυτές ε, θα χρησιμοποιηθούν και για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των πολιτικών που θα επιτρέψουν την χρήση των διαρθρωτικών μέσων κατά την επόμενη προγραμματική δημοσιονομική περίοδο. Και εμείς συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις οι οποίες ελπίζω να ολοκληρωθούν με κάθε μία από τα κράτη-μέλη το ταχύτερο δυνατόν έτσι ώστε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι προτεραιότητες αυτές θα συμπεριλάβουν και θα αντικατοπτρίζουν τις ειδικέ αναχώρα συστάσεις. Λοιπόν, ο στόχος ένταξης των Ρωμά λοιπόν θα συμπεριληφθεί στις εταιρικές αυτές ε, εταιρικής φύσεως συμφωνίες και θα αντικατοπτρίζεται στην σωστή κατανομή των πιστώσεων στα πλαίσια της χρήσης των διαφθορτικών ταμείων. Να μου επιτρέψετε παράλληλα να αναφερθώ τώρα στις συστάσεις προτάσεις μάλλον τις προτάσεις για συστάσεις του Συμβουλίου που υιοθέτησε τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της έκθεσης αξιολόγησης. Πρώτον, θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για την υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη την οποία επέδειξαν τα εθνικά σημεία συντονισμού Ρωμά από τις διάφορες χώρες μέλη και τις 14 χώρες που πήραν μέρος στην προπαρασκευαστική προσπάθεια. Γιατί ήταν σημαντική αυτή η προσπάθεια, μα διότι εμείς είχαμε σαν στόχο μέσω της υιοθέτηση της συγκεκριμένη προτάσεως ένα διπλό θα έλεγα επίπεδο πλαίσιο για τη συμπερίληψη και ένταξη των Ρωμά στον κοινωνικό και οικονομικό χώρο και δεύτερον θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχουν μπροστά τους οι χώρες και θα θέλαμε με τη σύσταση αυτή όχι μόνο να προσανατολίσουμε και να δώσουμε στα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μια σωστή γραμμή αλλά να στηρίξουμε και την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων αυτών σημείων συντονισμού αναχώρα. Επαναλαμβάνω, αυτά τα σημεία συντονισμού αναχώρα δεν έχουν την πολιτική στήριξη και τις αρμοδιότητες έτσι ώστε να φέρουν απρόσκοπτα εις πέρα στην αποστολή τους. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για τις προτάσεις αυτές για συστάσεις του Συμβουλίου. Καλύψαμε τα εξής θέματα υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων και μέτρων στόχων για την ίση μεταχείριση των Ρωμά στην πρόσβαση στην κατοικία, την ε, ιατρική φροντίδα, την εκπαίδευση, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας. Εφαρμογή των βασικών αρχών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των κοινοτικών αλλά και εθνικών πιστώσεων, που χρησιμοποιούνται για την ένταξη των Ρωμά, βασικά οριζόντια διαφθρωτικά μέσα όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προστασία των γυναικών και παιδιών Ρωμά. Σύμφωνα με το πακέτο που υιοθετήθηκε στις αρχές του χρόνου, το λεγόμενο πακέτο κοινωνικής επένδυσης. Επίσης και η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ηγετών των κοινοτήτων Ρωμά, διότι η αλλαγή θα γίνει και από μέσα και όχι μόνο από πάνω. Ε, η σωστή μεταφορά των εθνικών ανηλυμένων υποχρεώσεων σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό διότι έχουμε την αίσθηση και το είδαμε αυτό ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα και δεν είναι επαρκές να σχεδιάζει κανείς κάποιες σωστές πολιτικές σε επίπεδο κυβερνητικών κανόνων, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό οι πολιτικές αυτές να είναι ρεαλιστικές, να είναι εφαρμόσιμες και ε, όταν ερχόμαστε στα θέματα της εφαρμογής να υπάρχει δυνατότητά τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Να υπάρχει σωστή παρακολούθηση των εξελίξεων της εφαρμογής των πολιτικών Υπάρχει ένα μέσο αξιολόγησης μέσω ακριβώς των οδηγιών οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η ενίσχυση των πόρων που είναι διαθέσιμη για τα εθνικά σημεία συντονισμού Ρωμά και μορφές συνεργασίας ανάμεσα στις γειτονικές περιφέρειες, ανάμεσα στις τοπικές αρχές τις τοπικές κοινότητες που ε, δεν είναι βέβαια όμορες υποχρεωτικά αλλά παρόλα αυτά ε, είναι σαν παράδειγμα χώρες προέλευσης ή χώρες κατάληξης κάποιων ε, μετακινήσεων Ρωμά όταν οι Ρωμά ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη διακίνηση. Θα ήθελα λοιπόν για να κλείσω την παρουσίασή μου πλέον να πω ότι η πρόθεσή μας από εδώ και στο εξής είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τα Εθνικά Σημεία Συντονισμού Ρωμά, να συνεργαστούμε επίσης στενότερα με την κοινωνία των πολιτών, με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη-μέλη και με μια ολόκληρη σειρά διεθνών οργανισμών έτσι ώστε να προετοιμάσουμε ένα πλήρως αναπτυγμένο θα έλεγα πρόγραμμα αξιολόγησης στις αρχές του επόμενου χρόνου που θα μας δείξει ακριβώς την πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στους βασικούς τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατοικίας και πρόσβασης στη δημόσια υγεία. Μέχρι τώρα έχουμε αξιολογήσει τις εθνικές πολιτικές όπως έχουν καθοριστεί στα εθνικά αν θέλετε έγγραφα Έχουμε δει τι ακριβώς γίνεται με τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία καλούνται να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των πολιτικών αυτών. Είδαμε τις δυσκολίες και τα ελαττώματα των μέτρων αυτών, αλλά έχει φτάσει πλέον η στιγμή ή θα φτάσει ε, στις αρχές του 2014 για να αναφερθούμε και σε εσά και στο Συμβούλιο σε θεσμικό επίπεδο για την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί και για το τι δεν θα έχει επιτευχθεί στα πλαίσια της προσπάθειας εφαρμογής των πολιτικών αυτών και της συγκεκριμένης προόδου στον τομέα της παιδείας, επαναλαμβάνω, της κατοικίας κτλ. Αυτό είναι λοιπόν το επόμενο στάδιο, ο επόμενος στόχος και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να αναφερθούμε σε σας εκ νέου το αργότερο μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2014 είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια και ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζομπάν. Ντορντέα, εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τώρα αρχίζει η συζήτηση. Σημείωσα μερικά ονόματα συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Γκιόνς πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ για την έκθεση και την περίληψη Βλέπουμε όμως και με τη δική σας έκθεση ότι η κατάσταση είναι αρκετά απογοητευτική. Είπατε ότι δεν έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Εγώ το αντίθετο θα έλεγα. Δεν έχει επιτευχθεί τίποτα. Καμιά φορά η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ οι λόγοι και οι παράγοντες. Και επίσης αυτό που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη είναι η έλλειψη της πολιτικής βούλησης ή πάρα πολύ στοιχειώδη πολιτική βούληση για επένδυση σε αυτό το τομέα της ένταξης των Ρωμά. Και επίσης κάτι άλλο που βλέπουμε είναι επικοινωνία. Για παράδειγμα στην Ουγγαρία αναλώνονται στην επικοινωνία η κυβέρνηση ε, που και ο αρμόδιος ε, που είναι τώρα αρμόδιος για την ένταξη Ρωμά, στο παρελθόν ήταν αρμόδιος για τη στρατηγική επικοινωνία. Δεν έχει καμία σχέση με την ε, ένταξη των Ρωμά. Και παντού βλέπουμε την έλλειψη ε, στοιχείων αξιόπιστων, βασικών, που να μπορούμε να συγκρίνουμε και να μετρήσουμε τα επιτεύγματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με τον Οργανισμό Θεμελιδών Δικαιωμάτων που έχει βγάλει μια έκθεση που δείχνει πάνω κάτω την ίδια εικόνα, ότι δεν έχουμε την παραμικρή βελτίωση ε, στην κατάσταση του Ρωμά, ανά την Ευρώπη, παντού. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε και με άλλους διεθνείς οργανισμούς ε, που επενδύουν ε, στη συλλογή στοιχείων δεδομένων στην παρακολούθηση της κατάστασης του Ρωμά με μεμονωμένα προγράμματα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης ότι καμιά φορά βγάζουμε πολύ ωραία χαρτιά για στρατηγικές για την ένταξη των όνομα, αλλά η πραγματική νομοθεσία και η πραγματική πολιτική βαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παράδειγμα, μειώνεται το υποχρεωτικό ωραίο ε, ηλικία ε, για τη φύτη σε σχολεία στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, ή χρησιμοποιούνται ε, τα κονδύλια σε λάθος σκοπό όχι για την ένταξη των Ρωμά, αλλά για την ποινικοποίηση ορισμένων από αυτούς. Ε, είναι προσοχή λοιπόν αυτό που χρειάζεται στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων στο προσεχές πολιετές ε, πλαίσιο για να εξυπηρετεί πραγματικά την ένταξη των Ρωμά. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, στις συστάσεις του Συμβουλίου όταν αυτές ολοκληρωθούν, θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε σαφείς ως προς τις ευθύνες των κρατών μελών για την ισότητα της μη διακρίσης κτλ. Διότι παρόλο που έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, καμιά φορά φοβούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου όταν πρόκειται για τους Ρωμά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να συνεχίσουμε να πιέζουμε, να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε, να κοιτάμε την κατάσταση, να συλλέγουμε στοιχεία, βασικά στοιχεία, συγκρίσιμα στοιχεία, αξιόπιστα και με πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθούμε τι γίνεται στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, αν εξυπηρετούν πραγματικά αυτούς τους στόχους που έχουμε στα χαρτιά. Ακόμα και δεν υπάρχουν σαφείς δείκτες. Χρειάζεται πολύ μεγάλη πίεση για τα κράτη-μέλη για να μας ε, δίνουν αυτούς τους δείκτες και να συγκρίνουμε τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσομπάνου Ντορδέα, λέει η κυρία Βέμπερ, για την παρουσίαση. Δεν ε, αμφιβάλλω καθόλου ότι κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, χειριστεί το θέμα όσο γίνεται πιο σοβαρά, διότι σοβαρό είναι το θέμα. Ταυτόχρονα εγώ διατηρώ την αρχική μου άποψη. Με αυτό το πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές, για μένα δεν ήταν η σωστή η προσέγγισή μας. Και αυτό που χρειαζόμαστε ακόμα είναι ευρωπαϊκή στρατηγική, όχι εθνικές στρατηγικές. Μία ενιαία για όλα τα κράτη-μέλη. Και όχι ένα συντονισμό με εθνικά σημεία αναφοράς ή επαφής. είναι ευρέως γνωστό ότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την εφαρμογή καν της στρατηγικής ή των στρατηγικών αυτών, όπου υπάρχει, στα χαρτιά. Um, Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Εξ όσων κατάλαβα από αυτά που είπατε, ορισμένα από τα βήματα που θα ήθελε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον, ε, είναι αυτά που μας αναφέρεται. Αλλά εγώ έχω την εξής ερώτηση τώρα. Πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προθέσεις έχει για να αντιμετωπίσει ε, του, τις εκδιώξεις στο Ρωμά ε, από τη Γαλλία στην εποχή και του Σαρκοζή αλλά και τώρα του Ολάντ γιατί η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Προτίθεται να αναλάβει καμιά δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και τι σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον. Και επίσης θα πρέπει ίσως, έτσι για να διευρύνουμε το ερώτημα, να αναρωτηθούμε ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράδειγμα, ε, ως προς τη μελέτη ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το ζήτημα της ηθαγένειας. Η Ευρωπαϊκή ηθαγένεια... Είναι δυνατόν ε, σήμερα στην Ευρώπη ε, να βασίζεται στη φυλή, γιατί ε, υπάρχουν Ρωμά στους οποίους αρνούμαστε την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς σκέφτεται να το αντιμετωπίσει αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις δύο προλαλήσεις συναδέλφους και αυτό δεν σημαίνει κριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ακούγοντας τα όσα μας λέει ο κύριος Τσοπάνου, καταλήγουμε ότι έχουμε εκθέσεις, αναλύσεις, συστάσεις, παρακολουθήσεις, αλλά στην πράξη ουσιαστικά δεν έχει ακόμα αλλάξει σχεδόν τίποτα. Ακούσαμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Καμιά φορά λείπουν χρήματα, καμιά φορά λείπει εμπειρία για την ένταξη, αλλά ο βασικός πυρήνας και η ουσία είναι ότι συχνά ε, δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει προθυμία ουσιαστικά ένταξη στο Ρωμά με ε, τα αντίστοιχα σωστά ε, μέτρα. Και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, το είπε η κυρία Βέμπερ προηγουμένως. Τα χαρτιά δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Ορισμένα πράγματα φαίνονται ωραία στα χαρτιά, αλλά στην πράξη όχι. Παράδειγμα, ωραίο θα ήταν όλα τα παιδιά το Ρωμά να έχουν ε, πρόσβαση σε σχολεία, δικαίωμα να φοιτούν σε σχολεία, αλλά αν δεν τους διαθέτουν ε, οι δήμοι και οι κοινότητες ε, το μεταφερικό μέσο, τα λεωφορεία για να τα μεταφέρουν στα σχολεία, γιατί μένουν μακριά από τα σχολεία, τι να το κάνουν το δικαίωμα που έχουν πρόσβαση σε σχολείο. Το ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί πίεση και θέλει να φροντίσει ε, τα χρήματα όχι μόνο να ε, απορροφώνται αλλά να δαπανώνται και σωστά και να πιάνουν τόπο. Στη χώρα μου έχουμε κοινότητες ε, και οργανώσεις που σκέφτονται ε, να συνάψουν σχέσεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με άλλες κοινότητες σε άλλα κράτη-μέλη για να αναλάβουν αυτό το θέμα ένταξη στο Ρωμά και εκείνων που βρίσκονται στη Γερμανία, αλλά να τους βοηθήσουμε να εντάσσονται καλύτερα και στις ε, χώρες προέλευσης. Και εγώ διαρωτώ με, έχουν νόημα τέτοιες συνεργασίες εάν επιτόπου στις χώρες ε, προορισμού δεν υπάρχει πολιτική στήριξη για να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Δεν ξέρω, έχει ήδη κάποιες ιδέες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς μπορεί αυτό να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα. Ευχαριστώ. με euh, αυτό που είπε η κυρία Βέμπερ. Γιατί αυτό που είπε πρόκειται να προκαλέσει και άλλα σχόλια και άλλες παρεμβάσεις. Θα ήθελα να πω, ας πούμε στην κυρία Βέμπερ, ότι είμαι στη να όμιλο για τις ε, ε, επαναπροωθήσεις προς τη Γαλλία 400 ε, οι οποίοι έχουν ε, κρατηθεί κοντά στη Λιόν σε συνθήκες ουράς υγειονομικής που φαντάζεστε πώς είναι αξιοθρύνητες. Και Βεβαίως αυτοί είναι θύματα της μαφίας που δρά γύρω από το μεσχομένο και ανήλικοι που ζουν υπό τέτοιες συνθήκες. Οπότε και προσθέτουμε για αυτούς τους Ρωμά, την κατάσταση είναι εκρηκτική και λάβουμε υπόψη και τη γνώμη αυτών που μένουν εκεί γύρω. Φαντάζεστε κύριε Βέμπερ πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα μείνουν όσο έχουν. Αυτοί που είναι ο πάνω στον άλλο εκεί. Επομένως, τι γίνεται αυτές οι επαναπροωθήσεις μεταφράζονται διαφορετικά σε σχέση με την προηγουμένη κατάσταση υπό την προηγουμένη κυβέρνηση. Ναι, διότι ταυτόχρονα η τοπικές αρχές. Επίσης, οι περιφερειακές διοικητικές αρχές είναι υποχρεωμένες να τους ε, προστατεύσουν, να τους στεγάσουν. Κάποιοι άλλοι πάνε κάπου αλλού, όποτε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι πάνε εκεί, δεν φεύγουν και η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ταυτόχρονα δε. Πρόκειται εδώ για μια ορολογιακή βόμβα. Και θα πρέπει να θυμηθούμε το τι γινόταν επί προηγουμένης κυβερνήσεως σχετικά με το ίδιο θέμα. Ε, Επίση, καλά αυτό το λέω γενικότερα, λάβετε υπόψη το παράδοξο της κατάστασης στη Γαλλία, το ότι θα πρέπει να πάτε και να δείτε πόσο έχουν ενταχθεί στην γαλλική κοινωνία η Ρώμα. Είναι αυτή η πρωτοβουλία που λέγεται Αντάτου και τους έχει εντάξει αυτούς στην περιφέρεια της Λιών Και βλέπετε ότι υπάρχει λοιπόν στη Γαλλία όπως και αλλού, υπάρχει έντονη παραδοξότης, γιατί από τη μια μεριά έχουμε κάποια θετική πλευρά και από την άλλη μεριά τα πράγματα βρίσκονται σε εκρηκτικό σημείο για όλους. Και για αυτούς της χώρας υποδοχής και πολλές φορές φτάνουμε σε φαινόμενα βία τα οποία γίνονται όλο ένα και σοβαρότερα. Οπότε, γι' αυτό και εγώ τώρα αναρωτιέμαι για ποια στρατηγική μιλάμε, ευρωπαϊκή στρατηγική ή εθνική στρατηγική. Και εγώ μιλάμε σήμερα για ευρωπαϊκή στρατηγική, αναρωτιέμαι ακριβώς πού σημειώθηκε αυτή η πρόοδος που αναφέρεται στο κείμενο. Τι, ε, Τίποτα δεν κάναμε. Όλο τα ίδια και τα ίδια ακόμα και τελικά πάρα πολύ μικρά βήματα πρόοδο γίνανε τα τελευταία χρόνια. Κάτι άλλο επίση σαν προβληματισμός και διευκρινηση πρωτα πρώτα-πρώτα όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων νομίζω ότι ακόμα δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και θα ήθελα να μου διευκρινίσετε περαιτέρω εδώ Φελιππίν, ποια είναι η υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο των ε, ε, χωρών προέλευσης ή των χωρών ε, υποδοχής. Τι δυνατότητες υπάρχουν να υπάρξουν κάποιους προγράμματα, κάποιους κοινές, κοινοί κανόνες μεταξύ της χώρας προέλευσης και χώρας υποδοχής. Επίσης, τι γίνεται όσον αφορά την εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων διαφόρων φορέων, των ΡΟΜ, τη κοινωνία των πολιτών, των ΡΟΜ, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια βήματα πρόοδου όσον αφορά του. ΡΟΜ. Σας υπενθυμίζω, λέει ο Πρόεδρος, ότι πιέζει ο χρόνος. Διότι στις 10 θα έρθει ο διευθυντή της Υπηρεσία. Ε, υποστήριξης του ασύλου. Θα έρθει στις 10 ο επικεφαλής της ΕΑΣΟ. Οπότε έχουμε μείνει κάπως πίσω γιατί και άλλοι θέλουν το λόγο και θα πρέπει να τοποθετηθεί και η Γενική Διεύθυνση για το θέμα της ισότητας της Επιτροπής. Οπότε σας προτείνω οι υπόλοιποι να λάβουν το λόγο για ένα δίλεπτο. Κύριε Σίλτσεφ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Η έκθεση βεβαίως έχει συνταχθεί με τρόπο επαγγελματικό και υπεύθυνο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε για την ανάγκη να αλλάξουμε ορισμένα στοιχεία όλης της προσέγγισης του μοντέλου, του υποδείγματος που ακολουθούμε, θέλετε, του προτύπου. Η βάση τις όλες μας προσπάθειες πρέπει να αλλάξει. Διότι στις κοινότητες στο Ρωμά παρατηρούνται τώρα νέα φαινόμενα στην Ανατολική Ευρώπη. Επειδή αναφέρθηκε και η Βουλγαρία ε, μεταξύ των πέντε κρατών στο πρόγραμμα ε, με μεγάλη συγκέντρωση ε, πληθυσμό Ρωμά και ως Βούλγαρος μπορώ να πω ότι σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία σε 20 χρόνια η κυρίαρχη πληθυσμιακά κοινότητα στη Βουλγαρία θα είναι η Ρωμά. Από το 2007 στο πληθυσμό των νηπίων και των παιδιών ε, ε, πλειοψηφούν ήδη και σε 20 χρόνια όταν θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας θα είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα. Ορισμένες από τις χώρες αυτές όπως η Βουλγαρία ή κατά κύριο λόγο η Βουλγαρία τελικά μπορεί να γίνει κράτος Ρωμά. Δεύτερον, αυτή η αίσθηση και αναμενόμενη αύξηση πληθυσμιακή μεταξύ των Ρωμά δημιουργεί κάποιες προσδοκίες πολύ παραπλανητικές όσο και επικίνδυνες ε, που δημιουργεί προβλήματα επίσης και προκαλεί προβλήματα ως προς την ένταξή τους. Είναι μια νέα διαδικασία με νέες παραμέτρους και εμφανίζουν, αν θέλετε, μια απροθυμία να ενταχθούν, να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να ε, μπορούν να μιλούν ε, ε, τη γλώσσα της χώρας και να εντάσσονται στην κοινωνία. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν μεγαλύτερες διευκολύνσεις και παροχές και τελειώνω στην κοινότητα των Ρωμά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συζητούμε και για τις ευθύνες των ιδίων, των ηγετών τους και των ε, επικεφαλής. Θα πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι έχουν ίσα δικαιώματα αλλά και ίσες υποχρεώσεις για το μέλλον ε, των χωρών μας των ίδιων. Ευχαριστώ. Now, Mr. Bronze. Ο κύριος Μπρόνς, παρακαλώ σύντομος. Uh, I'm sure the of the... Ωραίες οι ε, ε, ε, προτάσεις ε, πολύ ευγενείς όλοι και πολύ ε, φιλικοί. Δεν θέλω να σας χαλάσω αυτή την καλή εικόνα, αλλά είναι λίγο παθητική η κατάσταση σήμερα των Ρωμά και είναι μάλλον εύγλωτη. Σίγουρα έχουν υποστεί δεινά και διώξει οι ανθρωπευτοί, αλλά σήμερα θα πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα για εκείνου. Του παρουσιάζουν σαν να είναι άβουλοι. Σαν κάποιοι που δεν μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο ζωή του, δεν μπορούν να αποφασίσουν τίποτα που να του αφορά καθόλου. Του λέγουν ότι θα πρέπει να σταματήσουν να ζουν με τον τρόπο που ζουν τώρα. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη χειραγώγηση για να μην πω τίποτα άλλο. Ε, γιατί να αλλάξουν τον τρόπο ζωής, γιατί ε, δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις καλώς, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν και στερεότυπα και να στιγματίζονται. Στερεότυπο σημαίνει ότι έχουμε μια εικόνα η οποία δεν αλλάζει, παραμένει η ίδια και στέρεη για πάντα το θέμα αναλάζουν οι άνθρωποι ή αν αλλάζουν οι εικόνες είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Βέβαια εμείς δεν το συζητάμε, αλλά... Στην καθομιλουμένη όταν ε, μιλούμε για στερεότυπο ε, εννοούμε ένα κλισέ, κάτι που περιγράφει γενικά και γενικεύει και χαρακτηρίζει τον κόσμο. Κανονικά οι γενικεύσεις είναι νοησίες. Αυτό που δεν θα πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόζουμε ε, έτσι, γενικούς χαρακτηρισμούς ε, για μια ομάδα ανθρώπων με λίγες εξαιρέσεις ή μικρές. Οι γενικεύσεις λοιπόν και χαρακτηρισμοί για τους Ρωμά είναι κάτι που γίνεται. Όχι μόνο από το κοινό αλλά και από αξιοσέβαστα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπω είναι και η Ευρωπόλ. Η Ευρωπόλ έχει εκδώσει ένα βιβλιαράκι την 1η Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Διακίνηση ανθρώπων, τράφικινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και αναφέρει τις εγκληματικές ομάδες που, και τους διακινητές ε, και με κατάλογο. Και ε, πρώτη θέση του καταλόγου είναι η Ρωμά. Και επίση κορίτσια και γυναίκες ε, Ρωμά αναφέρονται ως θύματα του τράφικη Και αν κανείς τα αγνοεί ε, ε, όλα αυτά και τα παραγνωρίζει, διονύζει τον κίνδυνο. Ο Βρετανικός τύπος παραπλανητικά περιγράφει Βουλγάρους και Ρουμάνους πολίτες και τους χαρακτηρίζει εκείνους που βαίνουν σε παραβατικές πράξεις, ε, στους δρόμους ε, της χώρας. Ε, δεν είναι Βούλγαροι και Ρουμάνοι, είναι Ρωμά περισσότεροι. Δεν, δίνω, δεν λύνονται τα προβλήματα όταν τα οροποιούμε και χρησιμοποιούμε ωραία γλώσσα και παραγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Κυρία Ματιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η στρατηγική την οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Ρωμά είναι κάτι το πάρα πολύ επενέσιμο, αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Οι Ρωμά έχουν προβλήματα ένταξης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε κάποιες χώρες έχει προχωρήσει η ένταξη, σε άλλες όχι, στις περισσότερες όχι. Ε, ο πληθυσμός αυτός έχει προβλήματα πολιτισμού λέει η κυρία Ματιέ ε, σε σχέση και με την εικόνα ε, που έχει η κοινή γνώμη. Ένας πληθυσμός που δεν επιτρέπει στα παιδιά να πηγαίνουν σε σχολείο μετά τα 12 ε, μόνο και μόνο γιατί τα κοριτσάκια πρέπει να παντρευτούν μετά τα 12, αυτό είναι πολύ σοβαρό και επίσης το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες εν πολλής. Οι πληθυσμοί αυτοί είναι σωστρεφείς και δεν μπορούν να ενταχθούν φυσικά με τους υπόλοιπους πληθυσμούς, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία βρίσκονται. Αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο δεν πρόκειται να ενταχθούν, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Έχω πάει στη Ρουμανία και είδαμε αρκετούς συναδέλφους το τι συμβαίνει και νομίζω ότι η έλλειψη εκπαίδευσης αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να συναντηθούν με τα υπόλοιπα παιδιά χάνονται για την κοινωνία, χάνονται για την κοινή γνώμη και δεν μπορούμε πάντα να λειτουργούμε με μια τέτοια εσωστρέφεια. Φυσικά τα κρατη μπορεί να δίδουν χρήματα για την ένταξή τους, αλλά τα προβλήματα θα παραμένουν γιατί δεν θέλουν να ενταχθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θέλουν να ενταχθούν. Και ό,τι και να κάνουμε έχω την αίσθηση αυτοί είναι οι οποίοι δεν εντάσσονται και αυτοί υποφέρουν βέβαια από αυτό δυστυχώς. Όταν δεν επιτρέπεται στις γυναίκες από τους συζύγους τους να πάνε στους γιατρούς είναι προφανές ότι δεν μπορεί να είναι ευτυχής. Άκουσα αυτά τα οποία είπατε ότι δεν άλλαξε η κατάσταση ανάμεσα στο Σαρκοζή και στον Ολάντ. Κοιτάξτε τι είπε η κυρία Γκυγιόμ, είπε ότι ζουν με έλλειψη καθαριότητας, το καλοκαίρι με φρικτή ζέστη και το χειμώνα με πάρα πολύ κρύο. Πώς το αντέχουν αυτό. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε προγράμματα ένταξης ε, για τους Βορειοαφρικανούς, τους Ασιάτες και τους ε, ε, Αφρικανούς γενικότερα. Αλλά οι Ρωμά δεν δέχονται τη βοήθεια, πρέπει να το ζητήσουν και αυτοί. Νομίζω ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ανεπαρκής, διότι δυστυχώς δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε γιατί δεν θέλουν να βοηθηθούν. Δύο λεπτά ο επόμενος ομιλητής. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία από ό,τι φαίνεται μακροημερεύουν και σε αυτήν εδώ την αίθουσα και διαρωτώ με αν πράγματι οι συνάδελφοι έχουν συναντήσει τους Ρωμά και έχουν συζητήσει μαζί τους. Κυρία Ματιέ, δεν αναφέρθηκα σε εσά αν θεωρείτε ότι σα αφορά αυτό που είπα δικό σας πρόβλημα. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει νομίζω που βρίσκονται τα προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι η πολιτική βούληση των κρατών μελών να εντάξουν τους πληθυσμούς αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών αυτών είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες και όχι σαν μετανάστες ανεξαρτήτως της επιθυμίας κάποιων. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο λοιπόν και όχι η ευρωπαϊκή στρατηγική γιατί ε, δεν υπάρχει θα έλεγα παρά ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό για εθνικές στρατηγικές. Αυτό το πλαίσιο είναι καλό και υπογραμμίζει την προβληματική που χαρακτηρίζει τους ε, πληθυσμούς αυτούς. Γιατί αυτοί οι πολίτες είναι θύματα τράφικινγκ, γιατί δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, όχι γιατί δεν το θέλουν, αλλά γιατί δεν τους δίνουμε τα μέσα. Πώς χρησιμοποιούνται λοιπόν τα ευρωπαϊκά ε, δινάρια και πώς ε, εμπλέκονται με σωστό τρόπο ή όχι η κοινωνία των πολιτών. Το παράδειγμα της Γαλλίας ε, είναι θα έλεγα ε, ενδεικτικό. Η κατάσταση δεν είναι ίδια σήμερα ε, με αυτή που ισχύει επί Σαρκοζή. Παρ' όλα αυτά όταν μιλάμε με τις ΜΚΟ μας λέγουν ότι οι συλλογικές Εξ όσοι συνεχίζονται πρόσφατα 200 διώχθησαν από τη Σεν Σεντενή. Ήταν ένας καταβλισμός σε τρία οικόπεδα. Ένα από αυτά ανήκε στη Δημαρχία του Μπομπινί που δεν ζήτησε να διωχθούν. Παρ' όλα αυτά πήγε η αστυνομία και τους έδιωξε παρότι δεν είχε ζητηθεί η εκδίωξή τους. Είχα πάει εκεί και χάρη στην αιμονή την πολιτική του τοπικού δήμαρχου οι πληθυσμοί αυτοί ξαναβρήκαν έναν χώρο για να εγκατασταθούν για να μην τρέχουν δεξιά-αριστερά. Οι υποχρεωτικές αυτές μετακινήσεις στη Γαλλία συνεχίζονται και δεν είναι παραδειγματική θα έλεγα η, ε, η κατάσταση στη Γαλλία. Υπάρχει ένας νομάρχης βέβαια που ασχολείται μόνο με αυτό αλλά αυτός ο νομάρχης διορίστηκε αλλά δεν έχει τα μέσα και οικονομικά και δεν υπάρχει και πολιτική βούληση για να βρει λύσεις. Αν ακούσει κανείς αυτά που είπε ο Υπουργός ε, Εσωτερικών της Γαλλίας, διαρωτάται πού βρίσκεται η Γαλλία σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι μια καλή βάση εκκίνησης. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά έχει εντάξει τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών στις θέσεις της. Αυτό είναι καλό γιατί μέχρι τώρα μέναμε μόνο στις κυβερνητικές θέσεις. Και τέλος είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί το θέμα των πραγματικών αξιολογήσεων της κατάστασης γιατί σε πολλές χώρες ε, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Είναι επίγον λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει το ρόλο του είναι επίγον να προχωρήσουμε σε μια επαναξιολόγηση των πιστώσεων που είναι διαθέσιμες, διότι γνωρίζουμε ότι ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η χρήση των πιστώσεων αυτών δεν είναι και σπουδαία. Λοιπόν, σύντομα θέλετε να απαντήσετε κύριε Τσομπάνου, Ντορντέα. Πάρα πολύ σύντομα σας παρακαλώ, διότι από χρόνο έχουμε πέσει λίγο έξω. και έχουμε και τον κύριο Φίσερ που περιμένει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, σύντομος θα είμαι. Καταρχά θα ήθελα να ε, προσκαλέσω το Κοινοβούλιο επ' ευκαιρία να εκφράσει με όποιο τρόπο θεωρεί σωστό διαδικαστικά την υποστήριξη ε, για την πρόταση για τις συστάσεις του Ιουνίου που ενέκρινε τον Ιούνιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάση το άρθρο 292 των συνθήκων και με τη νομική βάση ε, του άρθρου 19 παράγραφος 1 του, ε, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδικαστικά δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί αυτή η πρόταση προς έγκριση από κοινού ε, από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φρονούμε όμως και προσωπικά ε, πιστεύω ότι το ε, κατέδειξε και η σημερινή ένταση των συζητήσεων ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να μην παραγκονιστεί πολιτικά και να εκφράσει την άποψή του για τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στις στάσεις αυτές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις προτάσεις και τα σχόλιά σας και για τις επικρίσεις που εκφράστηκαν. Θα ήθελα να υπογραμμίσω παρόλα αυτά ότι εδώ πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για εθνικές στρατηγικές ένταξεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι μεν σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν καθοριστεί ήδη από το 2011. Αλλά μιλούμε ακόμα και για μίσο όπως είναι η στέγαση, η παιδεία ή ακόμα και η δημόσια υγεία η απασχόληση που δεν είναι κοινοτικές αρμοδιότητες, είναι κατεξοχήν εθνικές. Είναι ζητήματα των κρατών μελών, οπότε η ευθύνη είναι στα κράτη-μέλη για να χαράξουν και να εφαρμόζουν στη συνέχεια ε, τις εθνικές στρατηγικές. Είναι Εκεί η βασική ευθύνη σε σχέση με τα όσα μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διευθυντικά ταμεία διαθέτει πόρους οικονομικούς για την ε, άσκηση και εφαρμογή των, οικονομικών, των εθνικών πολιτικών. Συγγνώμη. Και όπως είπε μόλις η κυρία Βερζιά, είναι σημαντικό να απορροφώνται τα κονδύλια αυτά, αλλά με τη σωστή χρήση και να έχουν πρόσβαση όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και η κοινωνία των πολιτών όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως σας είπα προηγουμένω, έχουμε δρομολογήσει ένα πολιτικό μηχανισμό ε, που ορίζει κάποιους πολιτικούς στόχους και θα υπάρξει και ένας μηχανισμός στη συνέχεια για απορρόφηση των κονδυλίων όπου χρειάζονται. Αλλά υπάρχει επίσης ανάγκη να τα γνωρίζουν όλα αυτά οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακές και να αναγνωρίζουν και τα κράτη-μέλη τη πολιτική σημασία της ένταξης της πολιτικής αυτής, τις προτεραιότητές τους για την απορρόφηση των διαρθρωτικών πόρων την επόμενη επταετία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η πολιτική πίεση στα κράτη-μέλη. Εμείς από πλευράς της Κομισιόν θα το κάνουμε και θα το Υποβάλλουμε ξανά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όποτε χρειάζεται. Παρακαλούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το πράττει αυτό. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και με διεθνείς οργανισμούς και με ε, τις τοπικές αρχές ε, τους επόμενους μήνες για να εντοπίσουμε προγράμματα που μπορούν να εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο και να δείχνουν ε, το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουν στην κάθε χώρα οι τοπικές αρχές. Ε, τελειώνω. Πρόεδρε, με ένα ειδικό ζήτημα. Αυτό που ανέφερε η κυρία Βέμπερ για την κατάσταση στη Γαλλία, εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι μετά τον εντατικό διάλογο, και ξέρετε τι εννοώ λέγοντας εντατικό διάλογο που είχαμε το 2011 και το 2012 με τις γαλλικές αρχές, η γαλλική κυβέρνηση φθηγράμισε ε, την ομοθεσία της και την προσάρμοσε πλήρως στην οδηγία 38 του 2004 για την ελεύθερη διακίνηση. Είναι ειδικέ οι περιπτώσεις, τις γνωρίζουμε και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις και οι πρόνοιες της οδηγίας αυτής. Και οι ε, γαλλικές αρχές ε, συμμορφώνονται προς αυτή. Και σε περίπτωση που υπήρξαν εξώσεις ή εκδιώξεις ε, και αυτές ε, φέρονται ενώπιον της δικαιοσύνης για να αποφαίνεται ως προς το νόμιμο ή όχι. Και πολλές φορές και τα δικαστήρια απορρίπτουν αυτές τις αιτήσει. Ε, λειτουργεί λοιπόν ο νόμος, εφαρμόζεται και πέρσι εξεδόθηκε μία εγκύκλειο σχετική ε, ο πρόεδρος συντομεύεται παρακαλώ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσομπάνο. Ήταν ε, πάρα πολύ βασική αυτή η ζήτηση όσον αφορά την υλοποίηση των ε, στρατηγικών παρέμβαση για το Ρωμά και τώρα πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος γιατί θα πρέπει να πάμε στο σημείο παρελθόν 8 της στις όπω όπως είπαμε γιατί εδώ έχουμε καλέσει να συζητήσει μαζί μας στην Επιτροπή Λίμπε τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποστήριξης ε, του ασύλου. ΕΑΣΟ ονομάζεται, είναι ο κύριος Ρόμπερτ Βίσερ, καλώς ορίσατε κύριε και θα μας πείτε τα σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριότητας για το έτος 2012 όσον αφορά την κατάσταση που αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αφού κάνετε την εισηγησή σας θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής μας. και ε, έχω κάποια υποχρέωση, πρέπει να πάω κάπου άλλο και κάποια άλλη, αλλού για κάποια άλλη κοινοβουλία. θα με εγκαταστήσει κάποιος από τους, ή τις αντιπροέδρους. Ευθύς αμέσως για το λόγο κύριε Βίσσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Ήρθα σήμερα να σας παρουσιάσω την έκθεση για το 2012 που αφορά τις δραστηριότητες της ΕΑΣΟ. Και επίσης να σας πω τι ισχύει όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου να ε, δούμε πρώτα πρώτα σύντομα τι έγινε το 2012. Αλλά επίσης, μια που τώρα ε, έχουμε φτάσει σε πρώτη χρονιά του 2013, να δούμε τι γίνεται και το 2013. Το 2012 είχαμε 330.000 αιτήσει ασύλου στην Ευρώπη. Και, όπως μπορείτε να δείτε εδώ στην ε, επόμενη διαφάνεια, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει μια ελαφρά αύξηση εάν αυτά το συγκρίνουμε με το προηγούμενο χρόνο το 2011. Φέτος, επομένως, έχουμε ε, μια ελαφρά αύξηση ελαφρά, όχι πολύ μεγάλη. Όμως σταθερή να Η δε, δεύτερη κόκκινη γραμμή, χαμηλότερα, είναι οι νέε αιτήσει. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη, ότι με αυτές τις αιτήσει ε, φτιάχνουμε, από αυτές τις αιτήσεις, με βάση αυτών φτιάχνουμε τις ε, ε μας. Και η διαφορά μεταξύ των δύο είναι οι επαναλαμβανόμενες αιτήσει αυτών που επανέρχονται. Αυτό το οποίο μας, ε, απασχολεί είναι ότι ποιο είναι ο συνολικός αριθμός των ετούντων. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Είναι δηλαδή 10% αυτοί λιγότεροι από το σύνολο. Οι ετούντες το 2012 και ιδίω προέρχονται από Αφγανιστάν πρώτα-πρώτα, από Συρία που βέβαια ταχαίως ε, αυξάνονται και δεν χρειάζεται να σας πούμε γιατί. Οπότε έχουμε ε, κάποιο σύστημα εξέταση αυτών των αιτήσεων και επίσης από Δυτικά Βαλκάνια. Αν θεωρήσουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μία περιφέρεια. Κάτι που δεν γίνεται παντούτε, αλλά ομαδοποίησαμε τις χώρες αυτές. Και υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά που είναι κοινά στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Περιλαμβάνονται εδώ έξι χώρες. Ε, συνολικά λοιπόν η μεγαλύτερη ομάδα για πολλά χρόνια. Και φέτος. Όχι ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί αυτό διότι το πρώτο ημισή αυτής της χρονιάς είδαμε μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή στην Ισροή. Το Αφγανιστάν ακόμα είναι εδώ στον πίνακα, αλλά είναι στην τρίτη θέση. Η Συρία είπαμε ότι ανέβηκε και βέβαια είχαμε μεγάλη ανάγκη την περασμένη εβδομάδα. Αλλά στην πρώτη θέση φέτος έχουμε τη Ρωσία. Έχουμε κάποια ελαφρά αλλαγή στις τάσεις και βέβαια θεωρούμε ότι ακόμα είναι πρόημο για να εξαγάγουμε συμπεράσματα, αλλά στατιστικά βγάζουμε. Και κάτω-κάτω βλέπετε τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και είδατε όμως ότι και οι έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι κάτω από τη Ρωσία. Πάντως έχουν, έχει εποχιακό χαρακτήρα η εισρωή από τα Δυτικά Βαλκάνια. Και παραδοσιακά μέχρι τον Εύριο έχουμε άνοδο των αριθμών των ετούντων από τα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένω δεν χρειάζεται να είναι κανένα μάγο για να προβλέψει τι θα γίνει και φέτο επιβεβαιώστε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου είπαμε να καταπτυχθεί μια μελέτη, ε, να έχουμε κάποια συγκρισιμότητα όσο με τα Δυτικά Βαλκάνια. Και πρόκειται αυτό να στο παρουσιάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος του έτους να δείτε τι, τι, ποιες είναι οι μεταβλητές Τις διάφορες μεταβλητές λέγω να δείτε τις αλλαγές Βεβαίω, ε, προσέζει ενδιαφέρον η περίπτωση τη Συρία γιατί είναι θέμα καυτή επικαιρότητα και έχουμε εδώ μια ταχεία ραγδαία άνοδο των αριθμών και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα να προβλέψουμε οτιδήποτε για την εξέλιξη. Αλλά κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε εναρμονισμένη αντίδραση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η προστασία κατά κάποιο τρόπο παρέχεται στο 95 με 98% των ετούντων. Κάποιο είδους τέλο πάντων προστασία υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό επομένως το εξετάζουμε. Γιατί να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών στην προσέγγιση τους, μια που το τρόπο τέλεσμα είναι το ότι παρέχεται η αναγκαία προστασία. Επίσης, έχουμε συγκροτήσει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων, ειδικών, για να μπορούμε να έχουμε με ακρίβεια και καθημερινά επαφή με την επικαιρότητα, το τι γίνεται κάθε μέρα, τι αντιδράσεις υπάρχουν. Και είπαμε ότι προετοιμαζόμαστε για τυχόν εξελίξεις. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε δραματικές αλλαγές. Έχουμε τώρα 16 κράτη-μέλη, τα οποία έχουν εισρωή ατούντων από τη Συρία. Και σε αυτά τα 16 κράτη-μέλη η Συρία βρίσκεται στην πρώτη τριάδα όσον αφορά τους εισερχόμενους, τους ετούντες τέλος πάντων. Οι Γερμανοί και οι Σουηδία έχουν τους περισσότερους, αλλά και πέραν αυτών των χώρων βλέπουμε ότι και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουμε σύρου ετούντε. Ξαναγυρίζουμε για λίγο τώρα στην περσινή χρονιά και διαπιστώθηκε εκεί πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τα κράτη-μέλη, τα οποία επενδύουν στο σύστημα του ασύλου και ήδη προσπαθούν να ρυθμίσουν το του νέου πακέτου μέτρων. Βλέπουμε ότι υπάρχει ε, γενική, γενικός παράγον προστασία πάει στο 28% γιατί χειροτερεύσουν τα πράγματα σε κάποια μέρη του κόσμου, ε, στη Συρία, στο Μαλί, Φερρυπίνη. Αυτά, μια που πιέζει ο χρόνος και τώρα να δούμε κάτι άλλο. Τις δραστηριότητες της ε, ΕΑΣΟ. Κατάρτιση που είναι μια βασική μας δραστηριότητα όσον αφορά τη σύγκληση των ε, πρακτικών. Όλοι που ασκούνται με άσυλο θέλουμε να έχουν καταρτιστεί κατά τον ίδιο τρόπο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το ίδιο υλικό, ε, την ίδια ύλη να έχουν διδαχθεί και νομίζουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να φτάσουμε σε εναρμόνιση και συγκρότηση. ότι το 2012, 1,5 χρόνο, έχουμε καταρτήσει 2.481 υπαλλήλους. Πάρα πολύ σημαντικός αριθμός, γιατί έτσι ξεπεράσαμε κατά πολύ τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία είχαν τρέξει ε, τα προηγούμενα χρόνια για την κατάρτιση. Από αυτούς ε, κάποιοι ήταν Εκπαιδευτέ σε επίπεδο κρατών μελών. Οπότε εκπαιδεύσαμε τους εκπαιδευτέ. Είναι μία τη μεθόδου που χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης ε, είχαμε μια καταγραφή των ποιοτικών στοιχείων στα κρατημέλη και τα σχετικά του συστήματα και βοηθήσαμε στην βελτίωση. Επίσης έχουμε την πρακτική συνεργασία, τη συνεργασία σε πρακτικά θέματα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το τμήμα της δραστηριότητά μας αυτό. Το benchmarking και άλλα. Γιατί υπήρξε αρκετή ευελιξία να οργανώσουμε κάποια εργαστήρια, κάποιες συναντήσεις για τη Συρία, για την κατάσταση στη Ρωσία, όπου ε, φέτος είπαμε ότι είχαμε εξελίξεις και να έχουμε επίσης τέτοια επιχειρησιακά μέσα ε, σε επίπεδο συνεργασίας για πρακτικά θέματα. Τέλος, οι πληροφορίες όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των, ε, των ούτω ούτως ώστε να υπάρχει κάποια αξιολόγηση της κατάστασης στη χώρα προέλευσης και από αυτού έχουμε δύο μεγάλες σημαντικές εκθέσεις για το Αφγανιστάν και έχουμε και άλλες εκθέσεις ε, συντάξει, μικρότερες αλλά εξίσου μεγάλες σημασίες. Και έχουμε επίσης κάποια δίκτυα επιγραμμικά, τηλεφωνικά στο Ιντερνετ, για να συνδέονται οι εμπειρογνώμονε παντού και επίσης έχουμε και αυτή την διαδικτυακή πύλη που αποτελεί ε, σημείο ενημέρωσης για όλους την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε το σύστημα EPS για την έγκαιρη προειδοποίηση και προπαρασκευή. Πρόκειται για κάτι το οποίο βασίζεται και ορίζεται από την τρίτη συνθήκη του Δουβλίνου. Έτσι φτιάχνει αυτό το σύστημα. Και είπαμε αρχάς της φετικής χρονιάς θα αρχίσει η συλλογή των δεδομένων και εδώ και λίγες εβδομάδες έχουμε τα πρώτα δημόσια στοιχεία. Αυτό θα γίνεται σε ρυθμό τριμηνία, ούτω ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τα κρατημέλη για τις πολιτικές του ασύλου. Επίσης, παρακάτω, έχουμε την ειδική υποστήριξη για κάποιες καταστάσεις κατεπίγουσες που αξίζουν την προσοχή μας, πρώτα-πρώτα Ελλάς, Λουξεμβούργου, Σουηδία και Ιταλία. Ο καθένας είχε άλλες ανάγκες ε, και είχε διαφορετική υποστήριξη, αλλά για όλες αυτές τις χώρες αυτό ήταν αναγκαίο. Και ήταν η αποστολή μας να παράσουμε αυτή την υποστήριξη. Επίσης, εξωτερική διάσταση για πέρσι, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, ε, αυτό δεν ε, είναι το πρώτο σημείο ε, στη σειρά των δραστηριοτήτων, αλλά πάντως έγιναν κάποιες δραστηριότητες σχετικές, ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προσέξουμε ε, την Αφρική, οπότε ε, τώρα έχουμε επεκτείνει αυτή μας την δραστηριότητα και στην, για την Ιορδανία. Επίσης για τους ασυνοδεύτους λύκους, ανηλίκου, συγγνώμη, έχουμε αυτό το εγχειρίδιο όσον αφορά την αξιολόγηση της ηλικία, όσον αφορά την αναζήτηση της οικογένειας. Αυτό είναι μέτρο κατά του δουλεμπορίου ανθρώπων. Ε, συνεργασία επίσης με δικαστικές αρχές και δικαστήρια. Ε, επίση, έχουμε συνεργασία, αναπτύξη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την κοινωνία των πολιτών. Και παρακάτω έχουμε τις προτεραιότητες μας για το τι θα κάνουμε. Το 2014 ε, θα εστιάσουμε την προσοχή μας και το πλαίσιο το οποίο θα μας ε, καθορίζει θα είναι το, η νέα δέσμη μέτρων για το άσυλο. Και βεβαίως δεν μπορούμε παρά να σας ευχαριστήσουμε που ψηφίσατε και εγκρίνατε αυτό το θέμα γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα αναβαθμιστεί η πολιτική μας, θα πάμε από τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή στην εναρμόνιση, αυτό θα είναι τεράστιο βήμα προόδου, θα απαθετεί πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, πάρα πολύ προσοχή θα δοθεί στην υλοποίηση και επομένως και εμείς με τη σειρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτήν την διαδικασία. Τώρα, το δίκαιο στην πράξη. Διότι, όντα νομικό, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νομοθεσία και η νομοσχεδιαστική διαδικασία, αλλά αυτά θα πρέπει να μένουν νεκρό γράμμα και θα πρέπει να εφαρμόζονται και να μην εκπλαγείται, διότι πάλι βασικά θα εστιάσουμε την προσοχή μας εις την ε, κατάρτιση, στην ανάπτυξη ε, διαδικτυακών δικτύων και στην συνεργασία σε πρακτικά θέματα. Επίσης θα έχουμε ε, πάλι αυτό το σύστημα ε, της έγκαιρης προειδοποίησης και προπαρασκευής. Επίσης ε, θα πρέπει να αναμένεται την καταπαραγγελία ας το πούμε, ή ανάλογα με τις ανάγκες, υποστήριξη των κρατών μελών, όπως είπαμε και την Ιταλία, για να μπορέσει να εφαρμόσει τη δέσμη των μέτρων για το άσυλο και αυτά τα κρατημέλη να τα βοηθήσουμε ούτως ώστε να ε, διορθώσουν κάποια κακό κείμενα. Βεβαίως, όλα αυτά που είπαμε θα πρέπει να γίνουν με την ανάλογη πρικοδότηση. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Αυτά τα οποία προσδοκάται από την Ιάσο μπορεί να γίνει από συγκεκριμένα πρόσωπα. Και αυτοί πρόκειται επίσης να υποστηρίξουν την πολιτική σας. Αλλά εγκατακλείδη πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το έργο το οποίο επιτελούμε ως υπηρεσία η ανθρώπινη πόλη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Χρειάζεται να υπάρχει μια συνέχεια των δραστηριοτήτων όπως η έγκαιρη προειδοποίηση και αν υπάρχει εκεί πέρα κάποια τακτή ε, παρακολούθηση μπορούμε να παρακολουθούμε τις νέες τάσεις, τις αλλαγές αλλά αυτό απαιτεί ανθρώπινους πόρους, προσωπικό. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας και να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίσε. Καλημέρα σε όλους σας, ε, κύριε Νετφέλτ. Τρεις-τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Βίξτον πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ που ήρθατε και για την εξαιρετική σας ε, παρουσίαση. Κάθε φορά χαιρόμαστε ε, που έρχεστε να μας ενημερώνετε για ε, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Στα κράτη-μέλη ανησυχώ πολύ ε, και αναφέρεται αυτό και στην ετήσια έκθεση για τον κίνδυνο που έχουν κάποιοι να επιστρέφονται σε χώρες που δεν υπάρχουν εγγύησεις για την μη ε, επαναπροώθηση. Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και τι μπορούμε να κάνουμε για να τον αποφύγουμε ή να τον αποτρέπουμε. Παράδειγμα, καλύτερη παρακολούθηση, καλύτερος έλεγχος των επιστροφών και των αντιστοίχων διαδικασιών. Και επίση τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, τι τους συμβαίνει μετά την άφηξή τους. Γίνεται σεβαστή η αρχή της μη επαναπροώθησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την νέα έκθεση για την εποπτεία των εξωτερικών ε, θαλασσίων συνόρων που έχουμε εδώ εισηγητή τον κύριο Κοέγιο η υπηρεσία σας πώς μπορεί να υποστηρίξει και αυτή την προσπάθεια. Μαζί με εσά και πολλούς συναδέλφους εδώ παρόντες είμαι και εγώ πάρα πολύ περήφανη για το Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου και το θεωρώ μεγάλο επίτευγμα και όντως θα δώσει και ναι, καλύτερες διαδικασίες και καλύτερα πρότυπα και προδιαγραφές για τους ετούντες άσυλο. Τώρα όμως έρχομαστε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πρόκληση που είναι η εφαρμογή που ήδη αναφέρατε των ε, κανονισμών και των οδηγιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ τιμώ πολύ το ε, ρόλο του ΕΑΣΟ και χαίρομαι και για το νέο μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης στον κανονισμό Δουβλίνου που θα επιτρέψει καλύτερη παρακολούθηση σε όλα τα κράτη-μέλη και όλο το μέλλον. Μέχρι τώρα αντιμετωπίσατε εσείς καμιά δυσκολία ε, σε κάποιο κράτος μέλος για τις διαπραγματεύσεις ή για τη συνεργασία, με τι άλλο, ε, για αυτό το θέμα. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Το σύστημα είναι προσβάσιμο μόνο για πολίτες που έχουν φτάσει στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούν άσυλο επιτόπου. Με τη φυσική τους παρουσία δηλαδή, έχουν πατήσει έδαφος ε, κοινοτικό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να περάσουμε στο επόμενο βήμα, μια τρίτη φάση αν θέλετε του συστήματος, Είναι επικίνδυνο να φτάσει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανείς. Πολλοί πνίγονται στη Μεσόγειο. Η πρόεδρος διακόπτει, Μπορείτε να ολοκληρώνετε. Ναι, ναι, τελειώνω. Λοιπόν, εσείς πώς προβλέπετε την επόμενη φάση. Ε, να υπάρχει ένας νόμιμος τρόπος ασφαλής ε, να έχει κανείς πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει άσυλο, δηλαδή χωρίς τη φυσική του παρουσία. Και πώς προβλέπετε το άσυλο και την νόμιμη μετανάστευση να την ε, ε, καθιερώσουμε με νόμιμες ε, έλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω περιορισμένο χρόνο, ναι, ζητώ συγγνώμη λέει η Πρόεδρος, αλλά θα πρέπει να είστε όλοι λίγο πιο σύντομοι, έχουμε χρονικό πρόβλημα. Θα δώσω δύο λεπτά το πολύ σε κάθε μιλητή. Ο κύριος Φαντεκάμπ και μετά η κυρία Γιώτοβα, η κυρία Μέτσουλα, ο κύριος Μπρόνς, άλλος κανείς. Θέλει το λόγο. Όχι. Κλείνει ο κατάλογος. Ο κύριος Φαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Φίσερ για την έλευσή του εδώ και την παρουσίασή του. Ήταν πάρα πολύ σαφής και ε, εξαιρετική. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, για τη Συρία. Είναι τεράστιο έργο ε, και στο βαθμό που το θέλουμε να υποδεχθούμε όλους τους πρόσφυγες από τη Συρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχεδόν ανέφικτο. Εσείς έχετε τίποτα επαφές με την Τουρκία και με την Ιορδανία για να συνεννοηθούμε λίγο για τα ρεύματα προσφύγων ή ετούντων ασύλου και όλα τα τα προβλήματα. Υπάρχουν και χώρες πλούσιες όπως η Νορβηγία και η Ελβετία συγγνώμη, ε, που έχουν και κάποιο διεθνή ε, ρόλο. Εσείς συνεργάζεστε με αυτές. Ε, και δεύτερη ερώτηση αφορά το προσωπικό. Λέτε ότι χρειάζεστε βυρογνώμονες για το δίκαιο του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και τα συμβόλαια σας ε, είναι αρκετά μόνιμα. Από την άλλη λέτε θέλετε και έκτακτο προσωπικό για μικρό χρονικό διάστημα. Ε, πώς ε, το βλέπετε αυτό και για τη Ρωσία. Το πρώτο εξάμεινο λέτε του 2013 οι περισσότεροι τούντες άσυλο έρχονται από τη Ρωσία. Αναλύσατε και ποιοι είναι αυτοί και πώς. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ε, λόγω του Πούτιν που φεύγουν από τη Ρωσία και ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κρύβεται τίποτα άλλο από πίσω. Ευχαριστώ κυρία Γιώτοβα. <clears throat> Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή όχι μόνο για την πολύ καλή παρουσίαση που έκανε, αλλά και για το περιεχόμενο της παρουσίασης του. Δεν μπόρεσα να διαβάσω το σύνολο της προτινόμενης ε, από τον κύριο Βίσερ ε, παρουσίασης, αλλά βλέπουμε ότι τα πράγματα με τη Συρία μπορεί να χειροτερεύσουν και τίθεται εδώ το θέμα για την ικανότητα που έχουν οι χώρες ε, να χορηγούν άσυλο. Μία από τις χώρες που υφίστανται πιέσεις είναι η Βουλγαρία και η Ελλάδα φυσικά είναι στα εξωτερικά σύνορα. Έχει αυξηθεί το βάρος των αιτήσεων 46% ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς η, η Επιτροπή ε, μέσω του, της υπηρεσίας που ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια δεν μας έχει δώσει πολλές ε, δυνατότητες ελπίδας. Μας είπε ότι έχουν μειωθεί δραστικά τα ποσά για ανθρωπιστική βοήθεια η αρμόδια επίτροπος και είπε ότι για τέτοιου είδους βοήθεια δεν έχουν μείνει παρά μόνο 2 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι το θέμα των εξωτερικών συνόρων είναι ένα θέμα σοβαρό. Ε, είναι κάτι το οποίο κατά τη διάρκεια του χειμώνα μάλιστα η κατάσταση θα είναι πολύ πιο σοβαρή. Είπατε ότι θα βοηθήσετε χώρες σαν τη Βουλγαρία και την Ελλάδα και το υπενθυμίζω αυτό για την περίπτωση προσφύγων από τη Συρία. Μέτσουλα. Ευχαριστώ, Δ. Φίσερ. Διάβασα την ετήσια έκθεση και χαίρομαι γιατί βλέπω ότι λειτουργεί και ε, σωστά από τη βάση της στη Μάλτα. Ευχαριστώ επίσης και για την παραγωγική συνάντηση που είχαμε τον Ιούλιο. Είδα πώς δουλεύετε από πρώτο χέρι και δεν έχω αμφιβολία για το ότι αξίζεται να χρηματοδοτηθείτε σωστά για να λειτουργήσει σωστά ε, ε, το σύστημα. Ξέρουμε ότι η Μάλτα ε, αυτή τη στιγμή υποφέρει από την αυξημένη προσέλευση προσφύγων και δυστυχώς τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να ξεπεραστούν ορισμένες ενδογενείς δυσκολίες όπως το μέγεθος της χώρας, η πυκνότητα του πληθυσμού και γι' αυτό η αλληλεγγύη των υπολείπων χωρών είναι σημαντική. Με απογοήτευση είδα στη σελίδα 47 ότι από τους 217 που έτυχαν διεθνούς προστασίας που ζητήθηκαν από τη Μάλτα μόνο 14 ε, επανατοποθετήθηκαν σε άλλες χώρες μέσω του Γιουρίμα και οι υπόλοιποι μέσω άλλων ε, θα έλεγα τρόπων συνεργασίας. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτό. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και η ΕΑΣΟ πρέπει να επιβάλλει, θα έλεγα, στα κράτη-μέλη να μην ζητούν προϋποθέσεις και κριτήρια που είναι απόλυτα απίθανο να εκπληρωθούν. Θα πρέπει λοιπόν το ΙΑΣΟ να το πει αυτό. Έχει τη νομική δυνατότητα να προωθήσει την, ε, τη μετακίνηση ε, ετούντων άσυλο στην κάθε χώρα σε άλλες χώρες και θα πρέπει όλοι με δίκαιο τρόπο να μοιραστούν τις ευθύνες τους. Έχει ξεκινήσει ένα φόρουμ το οποίο ε, θα ε, ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Θα πάρετε το λόγο κύριε Φίσερ σε αυτό το φόρουμ και ελπίζω ότι θα πιέσετε έτσι ώστε να τοποθετηθούν περισσότεροι ετούντες από τη Μάλτα σε άλλες χώρες. Μπρόνς. Ε, θα πρέπει φυσικά τα δικαιώματα να γίνουν σεβαστά Μερικές φορές βέβαια γίνονται επίλεκτοι μετανάστες. Όταν κάποιοι κρυφίως πηγαίνουν σε μια χώρα και μετά ζητούν ε, άσυλο, ε, θα υπάρχουν αμφιβολίες βέβαια για την ειλικρίνεια των δηλώσεών τους. Όταν όμως ε, τέτοιου είδους αιτήσει δεν γίνονται θετικά δεκτές, παρόλα αυτά παραμένουν στις χώρες αυτές μέσω άλλων διαδικασιών και μπορεί να φτάσουν και τα 10 χρόνια. Κάποιοι που παράνομα μπαίνουν σε μια χώρα όταν ανακαλυφθούν ζητούν άσυλο είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ενθαρρύνει την παράνομη μετανάστευση και είναι η πραγματική αιτία των θανάτων των πνιγμών στη Μεσόγειο. Ξέρουμε κύριε Φίσερ τι γίνεται με τους πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και τη Συρία. Αν δεν είχαμε βέβαια πάει εκεί να κάνουμε πόλεμο θα είχαμε λιγότερους μετανάστες. Η εμφύλια διαμάχη Ενθαρρύνεται από μυστήριες χώρες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ και αυτό η επιτομή της δημοκρατίας η Σαουδική Αραβία. Και φυσικά και κάποιες δυτικές χώρες εμπλέκονται και θέλουν μάλιστα να πάρουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος. Όταν υποστηρίζουμε λοιπόν πολεμικές διαδικασίες να μην εκπλησόμεθα γιατί οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θέλουν να φύγουν. Ευχαριστώ κύριε Μπρος. Τελευταία η κυρία Κέλλερ ζήτησε να μιλήσει και μετά κλείνει ο κατάλογος και θα απαντήσει ο κύριο Φίσα. Παρακαλώ, κυρία Κέλλερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που έχασα την εισαγωγική παρουσίαση. Είχα άλλε ανελημμένε υποχρεώσει σε άλλε επιτροπέ. Δεν θα ρωτήσω τίποτα που σίγουρα θα έχετε απαντήσει. Απλώ να τονίσω και εξ ονόματο των Πρασίνων ότι Άσο κάνει εξαιρετική δουλειά τεράστια σημασία και θα πρέπει να είναι από του θεμελιώδει πυλώνε πολιτική ασύλου και αυτό να το τιμούμε αντίστοιχα και στον προπολογισμό. Σήμερα δυσανάλογα εστιάζουμε στο να επαναπροωθούμε κόσμο ή να ε, τον αποτρέπουμε από το να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθούμε εκείνους που πραγματικά έχουν τεράστια ανάγκη. Και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών είναι πάρα πολύ σημαντική εξίσου, αλλά δεν είναι κάτι που θα πρέπει να ζητούμε να το λύσει η ΆΣΟ. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το αναγνωρίσουν και να το ε, ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη σε εκείνους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους λόγω διώξεων, διωγμών, πολέμων, διαφόρων ε, αιτιών που δεν είναι εύκολο να αναφέρουμε τώρα εδώ εμείς. Θα πρέπει να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και η Άσο μπορεί να μας βοηθήσει και τα κράτη-μέλη να ε, στήσουν σωστά συστήματα ασύλου, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα και να ε, υπάρχει μια ασφαλής προστασία των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ. Πανέρχομαι στον κύριο Φίσερ για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Uh, Θα απαντήσω με τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις αυτή τη φορά. Η κυρία Βίξτομ, εξωτιμή βουλευτή, ρώτησε για τις επιστροφές και τι γίνεται μετά την επιστροφή των ανθρώπων αυτών. Ω προς την δυνατότητα μη επαναπροώθησης. Κοιτάξτε, η ίδια η ουσία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου είναι μέσω της ποιότητας της διαδικασίας αλλά και της απόφασης να ε, εγγυάται ότι η επιστροφή και ο κίνδυνος ε, πραγματικά μη επαναπροώθησης να ε, αποσοβείται. Βέβαια ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος και πολύ περίπλοκος και η, κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία είναι βασικό στοιχείο ακόμα. Και από τακτικής πλευράς η μόνη λογική λύση σε αυτό το θέμα είναι εξή. Να είναι εγγυημένη μη επαναπροώθηση, να ελέγχεται σε βάθος και να εξασφαλίζεται απολύτως καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ε, όταν είναι στο σύστημα ασύλου κάποιος και μόνο με αυτή την εγγύηση μπορεί να ζητήσει ε, την επιστροφή κάποιου και ε, εκούσια και ακούσια όταν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επαναπροώθησης. Οποιοδήποτε σύστημα παρακολούθησης, τώρα θέλετε ένα παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης, μπορεί να ακούγεται αυτό ευχάριστο ή συμπαθές, αλλά δεν μπορώ να το συλλάβω, έτσι, και εγώ είμαι επιχειρησιακός. Δεν μπορώ να φανταστώ καν πώς μπορεί να, να στηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Λοιπόν, ας επικεντρωθούμε στην ποιότητα της διαδικασίας του ασύλου στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του νέου συστήματος, του νέου πακέτου. Γίνονται μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Και έρχομαι και στο δεύτερο τώρα σκέλος της ερώτησής σας, η συνεργασία των κρατών μελών. Στον έλεγχο και παρακολούθηση των δυνατοτήτων των κρατών μελών πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής και στην ευτυχή κατάσταση να σας πω ότι η συνεργασία μας αυτή είναι πάρα πολύ θετική και αγαστή. Έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Βέβαια πάντα κάποιο θέλει περισσότερα, είναι διαδικασία. Ορισμένα στοιχεία ακόμα δεν τα συλλέγουν όλα τα κράτη-μέλη. Ε, δεν μπορούμε να ζητούμε στοιχεία τα οποία δεν συλλέγονται. Αλλά είναι πολύ ε, θετική κατά τα άλλα η στάση των κρατών μελών. Συνεργάζονται ε, στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Eurostat και τη Frontex και εμείς για να ε, αποφεύγονται οι επικαλύψεις. Γενικά όσο γίνεται το σύστημα αυτό λειτουργεί της ε, παρακολούθησης και της συνέχεια. Η τρίτη φάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έρθει κάποια στιγμή και αυτή. Ο νόμος εξελίσσεται όχι μόνο Εθνικό και διεθνή. η νομοθεσία είναι μια δυναμική διαδικασία και η πράξη και στον κόσμο της μετανάστευση και η πραγματικότητα ε, είναι μεταβαλλόμενη, οπότε θα χρειαστούν ε, μοιραία κάποιες ε, προσαρμογές. Δεν είναι δικό μου θέμα να την κινήσω αυτή την αλλαγή, είναι νομοθέτες που το κάνουν, αλλά μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία θέλετε προς την κατεύθυνση αυτή. κύριος ρώτησε για τη Συρία, ε, για τις δυνατότητες δράσης στην περιοχή, ε, αν το μεταφράζω σωστά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τώρα το πρώτο καθήκον της ΕΑΣΟ. Εμείς επικεντρωνόμαστε στις δυνατότητες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε απολύτως δίκιο. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δραστηριοποιούνται σε αυτή ε, την κατεύθυνση και είμαστε σε στενή επαφή μαζί τους για να αποφεύγουμε πράγματι και επικαλύψεις και δίπλο δουλειές και να ενημερωνόμαστε όσο γίνεται ε, καθώς και να τους ενημερώνουμε όσο γίνεται. Οι συνδεδεμένες χώρες, ε, Ελβετία και άλλες, συμμετέχουν και στις εργασίες της ΕΑΣΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι δεδομένη η συνεργασία και οι επαφές. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό μας μόνιμο και έκτακτο προσωρινό. Έχουμε υπαλλήλους ε, και των δύο κατηγοριών. Έχουμε διαφορετική ονοματολογία, αλλά ουσιαστικά περί αυτών πρόκειται. Έχουμε πολλούς ε, μονίμους και κάποιους περιορισμένους εκτάκτους υπαλλήλους προσωρινούς ε, που είναι απεσπασμένοι συνήθως εθνικοί εμπειρογνώμονες για καταστάσεις προσωρινού χαρακτήρα ή που χρειάζονται προσωρινή ε, ενασχόληση. Ε, Ρωσία, Δυτικά Βαλκάνια. Είχαμε προσλάβει πραγματικούς εμπειρογνώμονες εκτάκτως για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τη Ρωσία, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 9 μήνες, 12 και μετά θα επανέλθουν, είναι αποσπασμένοι, θα επιστρέψουν στις πρωτεύουσέ τους. Και εμείς θα κοινοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα των ερευνών. Έτσι εργάζονται και οι εκτακτοί και οι μόνιμοι υπάλληλοι μας. Γιατί η Ρωσία και αν φταίει ο Πούτιν. Δεν ξέρω αν είναι θέμα Πούτιν αλλά γνωρίζω ε, το μέγεθος της ε, κατάστασης. Η ροή έχει αυξηθεί. Είναι κυρίως Τσετσένοι ή κάποιοι που δηλώνουν Τσετσένοι. Ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία, αλλά η πλειονότητά τους δηλώνουν Τσετσένοι και μάλλον είναι και Τσετσένοι. Για τη Συρία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών. Το θεμέλιο του κοινού συστήματος ασύλου είναι ότι κάθε κράτος μέλος ε, είναι υπεύθυνο για το σύστημά του και για τις δυνατότητες που έχει. Έχει γίνει αυτή η ε, ε, επιλογή, δεν είναι δική μου επιλογή ούτε θα πρέπει να τη σχολιάσω εγώ. Πώς έχει το σύστημα ΕΑΣΟ. Σε ειδικέ περιπτώσεις μπορούμε να δίνουμε λύσεις αναπερίπτωση για να βελτιώνεται η δυνατότητα. Το έχουμε κάνει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις και Ιδιαίτερα για τις χώρες που αναφέρατε, ε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και ακούμε τα μελήματά τους. Αν υπάρχει πραγματικά επίγουσα έκτακτη κατάσταση, ε, δεν μπορεί κανείς να αναμένει από κανένα κράτος μέλος να είναι προετοιμασμένο για τελείως ε, διαφορετικούς αριθμούς αφήξεων. Έχουμε ένα σύστημα όμως που μπορεί πολύ γρήγορα να δώσει έκτακτη βοήθεια, επίγουσα, και προσωρινή επιπλέον δυνατότητα ε, στα κράτη-μέλη για τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας σας. Το μόνο που δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ βάσει του κανονισμού είναι να λάβουμε την ε, απόφαση για κάθε άτομο ξεχωριστά. Αυτό παραμένει ε, στα κράτη-μέλη ως αρμοδιότητα. Για τη Μάλτα. Τα γνωρίζω αυτά πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είστε σωστοί στην εκτίμησή σας, η ε, Γιορίμα Απορρόφησε λιγότερους και έχουν γίνει οι δράσεις μάλλον διμερώς παρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε μια μελέτη περσινή για τους λόγους, τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία, Γιορίμα 1, Γιορίμα 2 και λάβαμε υπόψη επίσης και εξετάσαμε τις διάφορες διμερείς συνεννοήσεις και συμφωνίες. Δεν σας θα έλεγα ότι είναι αποτυχία η όλη επιχείρηση, γιατί είναι μεγάλη αριθμή τα νούμερα. Βέβαια πάντα μπορεί να είναι περισσότεροι, αλλά έχουμε καταλήξει στο εξή συμπέρασμα. Από τα γεγονότα και τα στοιχεία, τα πραγματικά που βρήκαμε. Ότι Χρειάζονται βελτιώσεις. Υπάρχει δυνατότητα και χώρος και από πλευράς των χωρών υποδοχής mm. και από πλευράς ε, των χωρών ε, προέλευσης, των κρατών μελών δηλαδή που στέλνουν αυτούς ε, τους ετούντες άσυλο. Θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα αργότερα κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου mm. και θα δούμε τι επόμενα βήματα μπορούμε να κάνουμε. Δια τελευταίες ερωτήσεις του κυρίου Μπρόνς και της κυρίας Κέλλερ. Νομίζω ήταν δήλωση περισσότερο. Βεβαίως οι πόλεμοι προφανώς παράγουν μετανάστευση και λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ αυτό κατά πόσο η, δυτική, η πολιτική των δυτικών κρατών ε, ευνοεί ε, λόγω της συμμετοχής σε πολέμους, της πρώτης πολέμων, τέτοια φαινόμενα. Κυρία Κέλλα, σας ευχαριστώ πολύ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Μας ευχαριστεί να ακούμε πόσο ε, μας παρακολουθείτε, τις εργασίες μας, μας αρέσει αυτό και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όχι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την προσοχή σας. Ε, uh, ευχαριστώ κύριε Φίσερ. Τελειώνει και αυτό το θέμα στη μέση διάταξη και περνούμε στο επόμενο που είναι η εκθέση του κύριου Κλάς. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη αφορά την τροπολογία στην προσθήκη της απόφασης 2009-35 σχετικά με τον κατάλογο των τρίτων χωρών και τις οργανώσεις με τις οποίες θα συνάπτει συμφωνία η Ευρωπόλ. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ζήτησε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για το μέσο αυτό και γι' αυτό θα δώσω τους εκπροσώπους τώρα την δυνατότητα της νομικής υπηρεσία μάλλον να δυνατότητα να παρουσιάσουν την γνωμοδότησή τους και μετά θα έρθουμε στους εισηγητές. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Κύριος Καϊόλη. Σύντομα, θα μπορέσω να σας μεταφέρω την περίπλοκη νομική απάντηση στις τέσσερις ερωτήσεις τις οποίες έχετε θέσει για τον κατάλογο των τρίτων χωρών και οργανώσεων με τις οποίες η Ευρωπόλ θα συνάψει συμφωνίες. Ε, θα αλλάξει λοιπόν μέσω της απόφασης αυτής η απάντηση προσθέτοντας τέσσερα επιπλέον θα έλεγα υποκείμενα ε, στο συγκεκριμένο κείμενο. Καταρχάς, κοιτάξτε συνάδελφοι, αν θέλετε να συνεχίσετε τη συζητήση σας παρακαλώ εκτός εθούσης. Κύριε Καγιόλα συνεχίστε. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι ούτε η νομική βάση επί της οποίας βασίζεται η πρόταση αλλά ούτε και η διαδικασία ε, την οποία επέλεξε το Κοινοβούλιο δεν φαίνεται να είναι σωστές. Η πρόταση βασίζεται σε έναν αριθμό άρθρων από διαφορετικές αποφάσεις του Συμβουλίου, αλλά όχι σε ένα συγκεκριμένο άρθρο της συνθήκης. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια κατάσταση που δημιουργεί μια δευτερεύουσα νομική βάση. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια νομική βάση που δεν προβλέπεται από τις συνθήκες και την οποία όρισε το ίδιο το όργανο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη εκφραστεί αρνητικά για τη δημιουργία μιας δευτερευούσης νομικής βάσεως μετά τη δράση την οποία ανέλαβε δικαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η δευτερεύουσα νομική βάση ξεπερνά τις δυνατότητες που προβλέπει η συνθήκη και υπονομεύει την αρχή της θεσμικής ισορροπίας, ιδιοργανικής ισορροπίας. Η ε, γνωμοδότηση αν γίνει δεκτή θα βασιστεί στην δευτερεύουσα και μόνο νομική βάση και μπορεί να αμφισβητηθεί. Περαιτέρω η διαδικασία που επελέγει για την εμπλοκή του Κοινοβουλίου δεν είναι σωστή. Η απόφαση του Συμβουλίου για τον κατάλογο των τρίτων χωρών με τις οποίες θα συνάψει συμφωνίες είναι ένα μέτρο που εφαρμόζει την απόφαση για την Ευρωπόλ. Αυτή η αρχική απόφαση του Συμβουλίου προτείνεται και θα γίνει δεκτή μετά από την πλήρη θέση σε λειτουργία και ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας μέσω των εφαρμοστικών μέτρων και των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό απαιτείται έτσι ώστε να διευκρινιστεί. Αν ο κατάλογος αυτός και οι αλλαγές στον κατάλογο αυτό θα θεωρηθεί κατεξουσιοδότηση πράξη ή εφαρμοστικό μέτρο. Η εφαρμογή που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την απόφαση αυτή, την απόφαση Ευρωπόλ, είναι η κανονική νομοθετική διαδικασία. Είτε θα πρέπει να τροπολογηθεί η απόφαση Ευρωπόλ και να διευκρινιστεί αν θα γίνονται και με ποιο τρόπο αλλαγές ή να αλλάξει η απόφαση ευρωπολ και να συμπεριληφθεί στη νέα απόφαση ότι η Ευρωπόλ θα μπορέσει να συνάψει συμφωνίες με αυτές τις τέσσερις επιπλέον χώρες. Τώρα για τη θέση του Κοινοβουλίου για την αρχική πρόταση και αν η θέση αυτή του Κοινοβουλίου θα επηρεάσει τη δικαστική διαδικασία. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η άσκηση του δικαιώματος του Κοινοβουλίου να αναλάβει δικαστική ε, διαδικασία δεν είναι κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί από το Κοινοβούλιο στον έφετο χρόνο. Το δεύτερο αφορά τους κανόνες που θα εφαρμοστούν αν η νέα συμφωνία για την Ευρωπόλ θα τεθεί σε λειτουργία πριν ολοκληρωθούν οι υπογραφές όλων των επιμέρους ε, συμφωνιών με τις τρίτες χώρες. Βασιζόμαστε από τον κανονισμό του Ευρωπόλ, τον νέο κανονισμό, όταν εφαρμοστεί συνεπώς, δεν μπορεί η νομική γνωμοδότηση παρά να δώσει μια υποθετική, αν θέλετε, άποψη, διότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε την τελική απόφαση. Η απόφαση την οποία σας δίνουμε βασίζεται στον προτινόμενο κανονισμό ως έχει σήμερα. Εάν λοιπόν ο νέος αυτός κανονισμός τεθεί σε λειτουργία πριν την κατάληξη όλων των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες συνεργασίες, τότε τα άρθρα 31 και 77 του προτινόμενου κανονισμού παραμένουν τα ίδια και οι νέες συμφωνίες θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσει του νέου κανονισμού Ευρωπόλ. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το 2.18 ε, της συνθήκης και θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες προστασίας σχετικές με την προστασία της ιδιωτικότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Το τέταρτο θέμα αφορά τις προτινόμενες αλλαγές στο νέο κανονισμό Ευρωπόλ σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις κάτω από τις οποίες θα συναυθούν οι συμφωνίες αυτές με τρίτες χώρες. Θα πρέπει να καθοριστεί αν οι υπάρχουσες συμφωνίες παραβιάζουν τον νέο κανονισμό και χρήζουν επαναδιαπραγμάτευσης. Το άρθρο 73 παράγραφος 2 του προτινόμενου κανονισμού λέγει ότι η θέση σε ισχύ του κανονισμού Ευρωπόλ δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη νομική ισχύ των συμφωνιών που συνήθισαν από την Ευρωπόλ πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του προτινόμενου κανονισμού, η Ευρωπόλ μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε μια αρχή άλλης χώρας, τρίτης χώρας ή μιας διεθνούς οργανώσεως επί τη βάση της συμφωνίας συνεργασίας που έχει συναφεί ανάμεσα στην Ευρωπόλ και την τρίτη αυτή χώρα πριν από την ημερομηνία θέση σε εφαρμογή του νέου κανονισμού Ευρωπόλ. Ως εκ τούτου λοιπόν το κείμενο του προτινομένου κανονισμού ως έχει τώρα προτείνει ότι οι συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς δεν παραβιάζουν τον κανονισμό Ευρωπόλ και δεν απαιτούν εκ νέου διαπραγμάτευση. Αυτά είναι λοιπόν σύντομα τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε στα πλαίσια της γνωμοδότησής μας. Αν έχετε ερωτήσεις είμαστε στη διάθεσή σας. Εμείς ευχαριστούμε Κλάς. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σύντομος. Είναι μια πρόταση τώρα να υπάρχει δυνατότητα για την Ευρωπόλ να κάνει συμφωνίες με τη Βραζιλία, Γεωργία, Μεξικό και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα κράτη-μέλη το έχουν ζητήσει αυτό ορισμένα και πρόκειται για επιχειρησιακή συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή και προσωπικά δεδομένα θα ανταλλάσσονται με τις εν λόγω τρίτες χώρες. Και αυτή τη στιγμή η πρόταση αυτή ήρθε στα χέρια μας, είδαμε ότι υπάρχει ενδεχομένω ένα πρόβλημα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ταυτόχρονα μια πρόταση για ένα νέο κανονισμό της Ευρωπόλ ε, για τη διαδικασία ε, να μπορεί η Ευρωπόλ να συνάπτει ε, σχέσει και συμφωνίες με τρίτες χώρες. Οι σκιώδεις εισηγητές απευθύνθηκαν στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να γνωμοδοτήσει Όλες οι πολιτικές ομάδες το ζήτησαν που εκπροσωπούνται εδώ για να δούμε ποια είναι η νομική εγκυρότητα και η βάση. Μόλις ακούσαμε ε, τη σύνοψη της νομικής υπηρεσίας και της νομοδότησης Δεν μπορεί να εγκριθεί λοιπόν τυπικά βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται με το προηγούμενο ε, κανονισμό και την προηγούμενη συνθήκη πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός Ευρωπόλ πριν τις διαπραγματεύσεις για τις τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας, υπάρχει πρόβλημα εγκυρότητας. Πριν ολοκληρωθούν οι συμφωνίες αυτές δηλαδή. Θα πρέπει να ισχύει ο κανονισμός ε, για να ακολουθηθούν αυτές οι συμφωνίες και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι σοβαρό ε, το ζήτημα αυτό για τα δεδομένα και λόγω και των χωρών με τις οποίες συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες. Εγώ συμφωνώ με τη νομική μας υπηρεσία του Κοινοβουλίου και τη γνωμοδότησή της. Εγώ δεν θέλω καθόλου να αμφισβητήσω την ανάγκη να κάνουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Τα κράτη-μέλη θα έχουν τους λόγους τους και θεμητό είναι να το ζητούν. Αλλά ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητούμε πιο σαφή ε, ρύθμιση και νομοθεσία και κανονισμούς που να μην ε, ε, πυροδοτεί αμέσως νομικές συγκρούσεις. Γι' αυτό προτείνω να απορρίψουμε την πρόταση όπως έχει αυτή τη στιγμή σε περίπτωση που το εγκρίνει το Συμβούλιο δεν μας μένει άλλη επιλογή παρά να καλέσουμε την Ευρωπόλ να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις τρίτες αυτές χώρες ε, μέχρι να εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός της και να τεθεί σε ισχύ. Σας ευχαριστώ. Σαφέστατα κύριε Κλάστα, είπατε ευχαριστώ πολύ. τώρα θα ακούσουμε τους σκιώδες ηγητές, πρώτα πρώτα για το ΕΛΚ, την κυρία Χιμένες, η οποία εκπροσωπεί τον κύριο Ντίας Δεμέρα. Έχετε δύο λεπτά. Ε, gracias. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πολύ πιο σύντομη. Δεν θα χρειαστώ δύο λεπτά ε, στη θέση του κυρίου Ντεμέρα, του συναδέλφου, ο οποίος θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή, τον κύριο Κλάς, διότι ε, ε, ε, συνεφώνησαμε με λοιπόν όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι όλη αυτή η θέσπιση αυτού του, του κανονισμού της νομοθεσίας για την Europal πρόκειται να ολοκληρωθεί. Ο κ. Δίας Ντεμέρα είναι ο αρμόδιος ηγητής, οπότε θα ήθελα εξ ονοματός του να σας πω ότι εκείνος θεωρεί ότι είναι το πιο λογικό, το πιο σωστό να αναβληθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σχέση αυτής, οπότε για αυτό το λόγο ε, αυτά πρεσβεύει ε, ο εισηγητή μα. Σα ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χιμένε, γιατί σα τόσο σύντομοι. Ο κύριο Βάιντεν Χόλτσερ για, το, για του σοσιαλδημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ και εγώ με τον εισηγητή. Νομίζω ότι έχουν υποθεί τα πάντα ε, με σαφήνεια και εμεί ανέκαθεν ακούμε ότι ε, στον κανονισμό Ευρωπόλη είναι κάτι το οποίο μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα που να δυσκολεύει τα πράγματα και που δεν έχει και νόημα. Ε, που ε, υπάρχει και τέτοια περίπτωση συγκρούσεων. Και δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες, υπάρχει και άλλος κατάλογος για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και δεν ξέρω αν τα επίπεδα ασφαλείας και εγγύησης ε, ανταποκρίνονται σε αυτά που εμείς επιθυμούμε. Ευχαριστώ κύριε Βάινχολτσερ. Η κυρία Αλφάνο απουσιάζει. Η κυρία Γκρισμπέκ από πλευράς φιλελευθέρων δεν επιθυμεί να μιλήσει. Ο κύριος Ταβάρες, εξ των Πρασίνων, απουσιάζει από τους συντηρητικούς. ουδείς παρόν, η κυρία Βερζιά, εξ ονόματος ε, της Ενωτικής Αριστεράς. Ναι, λέει η κυρία Βερζιά. Θα σας το πω σύνομα όπως το και προηγούμενοι συνάδελφοι. Κατ' συμφωνώ με τον κύριο Κλά. Αλλά. Αλλά. Οπωσδήποτε τον ευχαριστώ για τη δουλειά του. Νομίζω ότι ομόφωνοι είμαστε όσον αφορά το ότι θα πρέπει να προσέξουμε για το θέμα. ο δεκατάλογος αυτών των χωρών είναι ε, πολυπίκυλος και όπως έχει σήμερα η κατάσταση γνωρίζουμε ότι κάθε συμφωνία που αφορά την ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει ε, να είναι θέμα που να το χειρίζεται κανεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά δηλαδή τον κατάλογο αυτών των χωρών. Έχουμε κάποιε χώρε οι οποίε δεν έχουν το ίδιο δικαϊκό σύστημα όπω και εμεί, οπότε και αυτό είναι ενισχυτικό και έχουμε πρόβλημα μέσα όσον αφορά τη νομική βάση και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Σας ευχαριστώ κυρία Φερζιά. Άλλοι συναδελφοί θέλουν τον λόγο. Όχι. Εγώ θα θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο ούτε άλλος από πλευρά της Προεδρίας του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευρά τη Προεδρίας να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, συζήτηση. Επίσης να σας αναφέρω ότι τώρα το Συμβούλιο έχει πει ποια θέλει ως νομική βάση. Και αυτό είπαμε θα μας απασχολήσει όσον αφορά τον οικονομισμό και είπαμε ότι θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οπότε και εμείς χαιρετίζουμε το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, καταλαβαίνει ποιε είναι οι λειτουργικέ και τις ανάγκες και φυσικά δεν μπορούμε παρά να ε, λάβουμε υπόψη την ανάγκη για προστασία των δεδομένων. Οπότε θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία μα διότι ούτε εμεί, ούτε εμεί θέλουμε κάποιο είδους νομικού φραγμού να τεθούν ε, εμπόδια στι κοινέ μα προσπάθειε. Ευχαριστούμε. Η πρόεδρο, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, όντως, αυτού του είδου η συνένεση είναι κάτι το σπάνιο. Κύριε Κλάς, θα θέλατε να υποβάλλετε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τους και για την ομοφωνία που είναι σπάνια όντως. Και θέλω να ευχαριστήσω και την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Η ημερομηνία για τις τροπολογίες, εάν κάποιο θέλει υποβάλει τροπολογίες, είναι 24 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 17 δεκάτου. Επομένω. ολοκληρώνουμε έτσι αυτό το σημείο και πάμε στο σημείο 10. Έλεγχος ε, εποπτεία των εξωτερικών θρασιών συνόρων στα πλαίσια τη επιχειρησιακή συνεργασία με το συντονισμό της, ε, του, του, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας και τη διαχείριση της ε, συνεργασία. Αυτή. αυτής. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι σαν να είναι βγαμμένο από των Monty Python. Τέλος πάντων. Ο κύριος Κοέλιο είναι ο εισηγητής. για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Έχετε το λόγο κύριε Πολιό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πρόκειται περί μεγάλου Όχι, όχι, δεν είναι έκθεση, είναι έγγραφο εργασία. Σύντομα να σα αναφέρω τα εξή. Πρώτα-πρώτα, κάτι που ήδη το γνωρίζουμε. Κατά την τελευταία δεκαετία, Όλοι στην περιοχή έχουν φυγεί από γεωπολιτικές και οικονομικές ε, ε, εξελίξεις. Οπότε και οδηγηθήκαμε σε πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια. Οπότε αυτό επέδρασε και στην ροή της διακίνησης των προσώπων, τα δε κράτη του Νότου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ε, κάποιων οι οποίοι προέρχονται από την περιοχή της Μεσογείου για να θέλουν να φύγουν, που φύγουν διώξεις, συγκρούσεις, πολέμους ή τουλάχιστον να, να ζητήσουν ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον και διάλεξαν τη θαλασσία οδό για να μπορέσουν να διασχίσουν τα σύνορα. Πάντως, το φαινόμενο αυτό ε, δεν ισχύει, δεν, γίνεται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, είναι σημαντικό. Οπότε η κατάσταση που προκύπτει αφορά κάποιο είδου. Ε, ...ΑΙΦΟΡ, βιώσιμη μας αντίδραση, να μπορέσουμε αυτούς που φύγονται κυρίως από αυτές τις αφήξεις από θάλασσα να τους υποστηρίξουμε. Η πρότασή μας, ε, η πρόταση της Κομισιόν είναι σταθμισμένη, έχει το ίδιο στόχο, όπως και μια άλλη παλαιότερη απόφαση. Μιλώ για την απόφαση του Συμβουλίου που την ακύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο νομικό μέσο νομοθέτημα να ισχύει στο διεθνέ δίκαιο και έτσι να μπορούμε να δούμε τι θα ισχύει από τα των μελών για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τις ε, καταθάλασσα επιχειρήσεις ε, υπό την αιγίδα της Frontex. Όμως θέλουμε να προχωρήσουμε παρακάτω γιατί έχουμε ε, μια παλιά απόφαση, κάποιες καθηγητές γραμμές για αποβίβαση, για διάσωση διοκομένων. Αυτά τα κείμενα τώρα να αποκτήσουν νομική δεσμευτική ίσχυ, να είναι άμεσα ε, εφαρμόσιμες και εκτελεστές στα κράτη-μέλη και έτσι να διέπονται όλες οι δηλαδή καταφέρας επιχειρήσεις της Frontex ή τόσο πάντων από το συνδυασμό της Frontex. Και έτσι να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στις επικρίσεις των επιχειρήσεων της Frontex για έρευνα και διάσωση. Όλοι συμφωνούμε, πιστεύω, ότι είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε περισσότερη σαφήνεια από νομικής πλευράς όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όσον αφορά την φύλαξη των θαλασσιών συνόρων, όσον αφορά την αποβίβαση των διασωθέντων, των, των διοκομμένων τέλο πάντων, αλλά όλα αυτά να γίνονται με τον σεβασμό της αρχής της μη επαναπρόθεσης για να σας παραπέμπω σε αυτά τα εγγραφή Εκεί προσπάθησα να αξιολογήσω το πώς έχει κατάσταση σήμερα, να δούμε τις νομικές εξελίξεις, τις βασικές πτυχές που θέλει να καλύψει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται επίσης να ετοιμάσω το σχέδιο της ε, εκθέσεως μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. και δίποτε προτάσεις τυχόν έχετε και όπως προείπα στην πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων χρειάζεται στενή συνεργασία για να μπορέσουμε να τηρήσουμε το σφιχτό διάγραμμα και έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι αυτή τη θητεία. Και σας πενθυμίζω ότι αν δεν καταφέρουμε να εγκρίνουμε ένα καινούριο κείμενο, τότε θα συνεχίσει να ισχύει η απόφαση του Συμβουλίου. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εργαστούμε ταχαίως και να συμβαστούμε με το Συμβούλιο. Σε ευχαριστώ. Αν κανείς είναι να τα βρει με το Συμβούλιο, αυτός εσείς είστε. Οπότε, για να δούμε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Προεδρία, εάν θέλουν μπορούν να λάβουν το λόγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. το λόγο ο Δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να προσθέσω. Εγώ νομίζω ότι από δική μας επόψεων τα έγγραφα εργασίας του εισηγητή είναι ακριβέστατα στην περιγραφή, θα έλεγα, της βάσης του θέματος. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Να επαναλάβω απλά ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. από πλευρά της Λιθουανική Προεδρίας, ο κύριος Ζιγκεβίτσιους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την άποψη της Λιθουανικής Προεδρίας για ένα σημαντικότατο θέμα. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι μία από τις βασικές προ... Προ... προτεραιότητες της Προεδρίας μας είναι η ουσιαστική προστασία και διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεισφέρει στο να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανοιχτή, αξιόπιστη και ασφαλή. Πιστεύουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε ότι η Λιθουανία έχει προγραμματίσει περισσότερες συναντήσεις του Frontex από ό,τι στο παρελθόν, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή πρόοδος. Η πρόταση κανονισμού για την επίβλεψη των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων στα πλαίσια της συντονιστικής δράσης του Frontex είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε τις αρμοδιότητες μας έτσι ώστε η απόφαση του δικαστηρίου να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν. Όπως γνωρίζετε, η εξέταση αυτής της προτινόμενης ρύθμισης έχει ήδη ξεκινήσει στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου κάτω από την Ιρλανδική Προεδρία. Η Λιθουανία θα συνεχίσει την προσπάθεια. Είχαμε και την προηγούμενη Τρίτη μια συνάντηση της ομάδας εργασίας για τα σύνορα που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα μόνο. Να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι πρώτες αντιδράσεις των εθνικών αντιπροσωπιών ήταν θετικές, αλλά είναι προφανές ότι για κάποια θέματα υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί ευαισθησίας από πλευράς των κρατών μελών. Εμείς θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση η οποία θα αντιπροσωπεύει τις θέσεις του Συμβουλίου γύρω από το ε, συγκεκριμένο ευαίσθητο θέμα. Κάποια συγκεκριμένα άρθρα ε, που δημιουργούν θέμα είναι το 9 και το 10. Δηλαδή οι ε, καταστάσεις ανάγκης, η έβρεση αγνοουμένων, και περαιτέρω συζητήσεις απαιτούνται για το εύρος της πρότασης και για τις δυνατότητες. Uh, European Parliament's rapporteur, first of all, I would like to thank Mr. Coelho for them and at the same time I would like to assure the committee θα πρέπει επίσης uh, οι δυνατότητες αυτές να λαμβάνουν υπόψη τη σωστή ενημέρωση την οποία, η οποία θα έχει προηγηθεί κατά τη διάρκεια της συνέχισης της εξέτασης της προτάσεως από πλευράς του Συμβουλίου, της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Thank you. Um, then on behalf of S&D, Mr. Weidenholzer. Σε ευχαριστώ. Ε. Θα ήθελα να πω ότι από κοινού ε, θα προχωρήσουμε σε μια καλή έκθεση με τον εισηγητή. Ε, νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να ε, συμφωνούμε και με μεγάλο ενδιαφέρον βλέπω και το έγγραφο εργασίες. Υπάρχουν μερικά σημεία που είναι για μένα πολύ σημαντικά η αρχή της μη επαναπροώθησης σαφέστατα να ισχύει και εδώ και να εφαρμόζεται κιόλα, να είναι ε, εφαρμόσιμη. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το εξή: Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να λαμβάνονται πολύ γρήγορα αποφάσεις και υπό μεγάλης πίεσης και στρες. Και θα πρέπει το, και το καθεστώς του κάθε προσώπου να ε, αξιολογείται σωστά ε, και είναι δύσκολο σε κατάσταση τέτοια ναι. πίεσης και αυξημένου άγχους. Και επίσης υπάρχουν και πρόσωπα ε, των οποίων δεν μπορεί να διαπιστωθεί άμεσα η ταυτότητα. Επίσης είναι σημαντικό ε, όσοι βρίσκονται σε ένα πλοίο τη στιγμή που αυτό συλλαμβάνεται θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Κάναμε μια αποστολή και είδαμε μια επιχείρηση Frontex στην περιοχή της Αλχεσίρας και θα πρέπει να καταλάβουμε πού υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες και χωρικά δηλαδή και τοπικά. από πλευρά ελέγχων είναι σημαντικό αυτό να γνωρίζουμε που διεξάγονται αυτές τις δραστηριότητες. Όταν κάποιο με ένα φουσκωτό σκάφο πάει από το Μαρόκο στην Ισπανία, ας πούμε, πρέπει να ξέρουμε ποιε είναι οι οδοί ε, και ο κάθε ενδιαφερόμενος ε, τη στιγμή που συλλαμβάνεται θα πρέπει να, να ξέρει, να γνωρίζει πού βρίσκεται, ε, πού κατευθύνεται. Αυτό είναι σημαντικό γενικότερα. Πάντω υπάρχει μεγάλη ομοφωνία. Αυτό φάνηκε άλλωστε και από τι συνεδρίε των σκιωδών εισηγητών. Η κυρία Βίξτρομ είναι επόμενη. Thank you very much. And I do indeed Ευχαριστώ πολύ και εγώ καλωσορίζω ε, το έγγραφο εργασία του εισηγητού μα, του κυρίου Κόγιο. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σας πω ότι σέβομαι και εκτιμώ πολύ την προθυμία σας να εργαστείτε με ένα αρκετά σφιχτό χρονοδιάγραμμα για να το εγκρίνουμε το συντομότερο και είμαι πρόθυμη και εγώ να συνεισφέρω προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν θα πω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, μερικά μελήματα που έχω να σας αναφέρω και ανησυχίε. Η αρχή της μη επαναπροώθησης θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι καλύπτει τους πάντες, όχι μόνο πρόσφυγες και τούντες άσυλο και να γίνεται σεβαστή ανα πάσα στιγμή. Δεν μπορεί να υπάρχει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία εμπλό ε, ε, ούτε ε, όταν είναι σε κατάσταση κρίσης ή αποβίβαση των ενδιαφερομένων και σε κατάσταση μεγάλου άγχους και πίεσης. Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται πάντα σεβαστή. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε συλλογικές αναχαιτήσεις ή επαναπροωθήσεις στη θάλασσα. Συμβαίνει αυτό και πρέπει να το ξέρουμε σήμερα η ε, πρόταση έχει ήδη καθυστερήσει για πολλούς λόγους όπως γνωρίζουμε και προσωπικά ανησυχώ για διάφορες φήμες που κυκλοφορούν ότι το Συμβούλιο και η Προεδρία δεν είναι αρκετά φιλόδοξοι ως προς το πρόγραμμά τους και το χρονοδιάγραμμα για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να ασφάλω, αλλά έχω τους φόβους μου. και πάλι χρειάζεται να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και ελπίζω η Προεδρία και το Συμβούλιο τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ε, φροντίσουν να προχωρήσουμε. Το Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο και ο εισηγητής πραγματικά βιάζεται ε, να τελειώνει γρήγορα αυτό το θέμα. Τώρα σε εσά εναπόκειται. Το Κοινοβούλιο κάνει τη δουλειά. Θα πρέπει και εσείς να δείξετε ακριβώς την ίδια ε, προθυμία και σας εκλυπαρώ. Η κυρία Μπέκ που είναι σκιώδης εισηγήτρια, μάλλον γιατί είναι συντάκτης γνωμοδότης στην Επιτροπή Μεταφορών. Συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε μικρόφωνο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, συμμερίζομαι τις θετικές απόψεις που έχουν απέναντι στις ε, προτινόμενες ε, ε, θέσεις του κυρίου Κοέλιο. Στα πλαίσια τώρα της νομοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αναφερόμαστε στα θέματα έρευνας, διάσωσης και συντονισμού των διαδικασιών αυτών. Θα σας παρουσιάσω τους δύο βασικούς άξονες της Επιτροπής Μεταφορών που θα ψηφιστούν στις 17 ε, Σεπτεμβρίου. Καταρχάς, ε, η επιμόρφωση των ε, των λιμενικών και εδώ σε σχέση με τις συλλήψεις ε, εν Θα πρέπει οι ρήτρε που θα ισχύσουν να είναι συμβατές με αυτές οι οποίες υπάρχουν στο πρωτόκολλο ε, που αφορά το τράφικινγκ ε, με άλλους τρόπους επίγειους και αεροπορικούς. Αυτό είναι κάτι το που αφορά την ασφάλεια, την ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών και επίσης την ασφάλεια του σκάφους ε, του ιδίου. Σχετικά με την κατάρτιση λοιπόν τώρα των λιμενικών και των συνοριοφυλάκων αν θέλετε, η κατάρτισή τους αυτή θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και της νομικής κατάρτισης που προβλέπεται. Πρέπει με πρακτικό τρόπο να γνωρίζουν επίσης ε, το πώς θα βοηθήσουν Ε, τα πρόσωπα τα οποία είτε συλλαμβάνουν είτε διασώζουν. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε ε, στις ανάγκες που υπάρχουν σε ανθρωπιστικό επίπεδο να έχουν στη διάθεσή τους τα σκάφη αυτά τα περιπολικά τα απαιτούμενα ιατρικά φαρμακευτικά μέσα, να υπάρχει σωστή δυνατότητα συντονισμού και αν είναι δυνατόν, αν και αυτό είναι πιο δύσκολο, να υπάρχει και ιατρικό προσωπικό εμπλό. Λοιπόν, αυτά. Σχετικά τώρα με την συνεργασία, θα έλεγα ότι έχει σημασία να αυξήσουμε τα επίπεδα συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνουμε εύκολα βέβαια, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες που εμπλέκονται ε, στον έλεγχο των θαλασσίων μεταφορών. Και αυτό προτείνεται πολύ τακτικά στην Επιτροπή Μεταφορών γύρω από την ολοκληρωμένη πολιτική θαλασσίων μεταφορών. Θα πρέπει να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων επίβλεψης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια ε, ε, των θαλασσίων μεταφορών. Να μην πολλαπλασιάζουμε τα μέσα, αλλά να χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα μέσα και για την προστασία ε, των υποψηφίων μεταναστών. Είμαι πεπισμένη έτσι ότι οι δράσεις που θα αναλάβουν οι αρχές αυτές θα έχουν λιγότερο κόστος, μικρότερο κόστος και ακριβώς έτσι θα μπορέσουμε να ενημερωνόμεθα σωστά και ο ρόλος αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει να ρυθμιστεί καλύτερα, να περιγραφεί καλύτερα στον κανονισμό. Λοιπόν, χοντρικά αυτά είχα να σας πω, λέει η κυρία Γκρίσβεκ, συγγνώμη αν μακρηγόρησα αυτά σχετικά με τη διάσταση των μεταφόρων που είναι μια ειδική διάσταση αλλά και συμπληρωματική των εργασιών μας. Ευχαριστούμε κύριε Γκρίσμπερ. Κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εργασία αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί νομίζω ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ φιλόδοξη είναι μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Για μένα το βασικό θέμα είναι πώς αυτές οι καλές προθέσεις, ε, αυτά τα ωραία λόγια να γίνουν πράξη, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε σε κάθε περίπτωση ε, και να υπάρξουν εγγύσεις για τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα όλων στις δύσκολες συνθήκες, στις διάσωσες, πάνω σε μια σχεδία, πάνω σε ένα σκάφο. Οπότε και εγώ θα ήθελα να διεκπαιρεωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα το θέμα και επίσης ε, ακόμη έχουμε κάποιες ιδέες που μπορούμε να προσθέσουμε στο κείμενο όπως ας πούμε το θέμα του ότι οι υπάλληλοι ε, θα πρέπει να είναι πάνω στο σκάβο τόσο να μπορέσουν να ε, εκτιμήσουν, να αξιολογήσουν τι γίνεται. Και επίσης υπάρχουν ότι τα δικαιώματά τους και σχέση με τη μήνυ παραπρόθεση θα πρέπει να, να, να προστατεύονται από κάποιες εγγυήσεις άσχετα με το ποιο επιλαμβάνεται τις καταστάσεις επίσης θα και χρειάζεται και κατάρτιση για να δούμε πώς θα μπορούμε να παράσχουμε αυτές τις ε, ε, αυτές τις εγγύσεις για αυτούς που βρίσκονται στο σκάφος πως ε, θα μπορέσουμε να τηρήσουμε επίση και την κόκκινη γραμμή δηλαδή το ότι θα πρέπει να ισχύει πάνω απ' όλα η σωτηρία ανθρωπίνων ζώων κατά θάλασσα. Αλλιώς δεν έχει νόημα ε, η ίδια η Frontex. Τέλος πάντων, ε, όλα αυτά αποτελούν μια σωστή βάση, αλλά να δούμε πώς θα βεβαιωθούμε ότι αυτά τα δικαιώματα θα ισχύουν υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Και δεν είναι εύκολο γιατί κάθε περίπτωση εδώ είναι διαφορετική. Αλλά ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον μια που αυτό θα ε, φέρει τη διαφορά όσον αφορά την προστασία ε, αυτών των προσώπων σε συνθήκες αυτές της κατά θάλασσα. Κύριε Γιακολίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το συγκεκριμένο θέμα αγαπητέ Κάρλος είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα σε μια δραματική στιγμή θα έλεγα. Μιλάμε για την επίβλεψη των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων σε μια πολύ δύσκολη φάση, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο θάλασσα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έγγραφο εργασίας του κ. Κοέλιο είναι συμβατό με τις απαιτήσεις που υπάρχουν για την προστασία των προσώπων των μεταναστών. Είναι βασικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμοστούν στα πλαίσια του εγγράφου αυτού, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν και θα πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν μέσω της αυξανόμενης κυκλικότητας των πληροφοριών η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας μας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε εκ νέου, ιδιαίτερα την έρευνα και διάσωση στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι αλήθεια ότι ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή ε, σύρων ε, είναι ήδη πρόσφυγες γιατί ζουν σε περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα μέσα στον τελευταίο μήνα ήρθαν 3.500 Σύριοι στη Σικελία μόνο. Και σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει και στη Λιβύη, στην Αίγυπτο κτλ. Πέραν των 35.000 προσφύγων των τελευταίων δύο καλοκαιριών, στην Ιταλία, στη Μάλτα, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, Υπήρξαν και άλλοι συνάδελφοι που επισκέφθηκαν τον προηγούμενο μήνα στην Ισπανία και της υπηρεσίας Frontex μέσω της νέας εντολής την οποία του προσδώσαμε εδώ και λίγα χρόνια. Λοιπόν, εμείς ε, υπενθυμίζουμε ότι τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νότο της Ευρώπης ε, ξέρουμε τι συμβαίνουν στη Λαμπεντούσα Ξέρουμε ότι μιλάμε για την περίοδο μετά τη σύμφωση της Στοκχόλμης. Ε, ελπίζουμε ότι όπως είπε και ο Κάρλος η συμβιβαστική λύση την οποία θα καταλήξουμε να είναι του καλύτερου επίπεδου που μπορεί να υπάρξει αλλά να λάβουμε υπόψη μας την ειδική κατάσταση η οποία καλεί τη χρήση ειδικών μέτρων για τη Μεσόγειο. Πιστεύω λοιπόν όλα αυτά να ληφθούν σοβαρά υπόψη όταν ε, οι καταστάσεις ε, το επιτρέπουν. Άκουσα και αυτό που είπε ο, η κυρία Μάλστρομ και ξέρουμε όταν ε, ένα σκάφος το οποίο ήταν έτοιμο να βυθιστεί σώθηκε από τους κατοίκους ε, ενός χωριού στη Σικελία που δημιούργησε μια ανθρώπινη αλυσίδα και χέρι με χέρι βοήθησαν 200 άτομα ε, να ε, φτάσουν στην ασφάλεια. Λοιπόν, γίνεται κάθε προσπάθεια, απαιτούνται όμως και τα κατάλληλα μέτρα. Ευχαριστώ. Πριν επανέλθουμε στον εισηγητή, κύριε Βερζιά, τελευταία ομιλήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ φοβούμαι ότι θα είμαι λιγότερο συνενετική σε αυτή την παρέμβαση από ό,τι στην προηγούμενη μου. Κρίμα που τα θέματα μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα βλέπουμε κατακαιρματισμένα χωρίς να έχουμε τη συνολική εικόνα του προβλήματος. Πολύ δε περισσότερο όταν βλέπουμε τα αριθμητικά στοιχεία είναι λιγότεροι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ τα γνωρίζω πολύ καλά διότι η δική μου χώρα που ήταν από τις χώρες που δεχόταν τους περισσότερους μετανάστες σήμερα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο του ΟΣΑ μάλιστα, το μέσο όρο. Τίστε το ερώτημα γιατί αυξάνεται η πίεση στις χώρες του Νότου, γιατί όντως αυξάνεται η πίεση στις χώρες του Νότου. Θα έλεγα ότι αυτό είναι απόρρια δύο φαινομένων. Πρώτον, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας η ευρωπαϊκή νομοθεσία ξέρουμε ποια είναι, Δουβλίνο 2 που είναι η οδηγία του έσχους και επίσης συνέπεια της εθνικής εκάστοτε νομοθεσίας που είναι όλο και πιο περιοριστική και αυστηρή. Αν δεν έχουμε αυτή τη συνολική θεώρηση πάντα θα επικεντρωνόμαστε ε, στα επιμέρους θα βλέπουμε μικρές ψηφίδες χωρίς να έχουμε το σύνολο του ψηφιδωτού ε, για την πραγματικότητα του προβλήματος όπως ακριβώς έχει σήμερα. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να φέρω στη συζήτηση ότι δεν θα πρέπει ε, να θεωρούμε κάτι τετριμένο αυτό το θέμα της μετανάστευσης μπανάλ. Κατανοώ τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια άλλη χώρα. Δεν είναι αποσπασμένη η στάση και ε, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ιουκοσλαβία δεν ήταν καθόλου ε, αντίστοιχη με την Αραβική Άνοιξη. Ούτε σήμερα είναι η ίδια απέναντι ε, στους πληθυσμούς της Συρίας σε σχέση με κάποιους που έρχονταν από την Τινησία ή την Αίγυπτο. Και εγώ χαίρομαι που εχθές ανακοίνησε η Σουηδία ότι ε, από τις 14.000 σύρους έχει ε, τακτοποιήσει 8.000 σύρους. Γιατί για να είσαι σύρος πρέπει να, είσαι έχεις μεγάλο κουράγιο και στένος και θάρρος να φτάσεις στη Σουηδία για να σε αναγνωρίσει η Σουηδία με αυτό το καθεστώς. Και ελπίζω και άλλες χώρες να δώσουν το παράδειγμα αντί να βγάζουν ωραίους λόγους. Και προσπαθώ να ξεχάσω και τη στάση της Γαλλίας σε αυτό το θέμα που μου φαίνεται αρκετά ε, σουρεαλιστική. Τελευταίο, η διάσωση στη θάλασσα. Πώς να το πω. Δεν βρίσκω και τα λόγια μου. Είναι αρκετά τρομακτικό αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε ε, και προσπαθούν κάποιοι να πιέσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με, περί πρόκειται. Τελειώνω, Πρόεδρε θέλουν να υποχρεώσουν τα κράτη-μέλη να σέβονται, λέει, τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Η θαλασσία διάσωση είναι διεθνής υποχρέωση. Και τι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία για να υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη να σέβονται τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι μας καλά θα κάνανε, τώρα που θα πάνε τους δώσουν και το βραβείο των Αμπελιρίνης, να τα ξανασκεφτούν όλα αυτά και να έχουν στάση λίγο πιο σωστή όταν πρόκειται να σεβόμαστε το δικαίωμα στη ζωή που είναι το πρώτο από όλα τα βασικά και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Και τώρα ο εισηγητής μας για να κλείσει παρακαλώ κύριε Κοέγια. Πρόεδρε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους ε, ε, οι οποίοι έλαβαν το λόγο, όλους τους συναδέλφους και θα μπορέσω να λάβω υπόψη όλα όσα πρότεινα. Μέχρι τα τέλη του μηνός θα έχω ολοκληρώσει. Κατοπίν δε. αρχίσει ο τριμερής διαδρός με το Σύμβουλο για να δούμε κατά πόσο υπάρχει περιθώριο για συμβασμό ιού. Ε, ναι, άκουσα την κυρία Βίξτο που είπε ότι δεν είναι και τόσο βεβαία για το ότι το Συμβούλιο προτίθεται τόσο πολύ όσο εμεί να εγκρίνει το νέο κείμενο. Ελπίζω ότι αυτό το οποίο είπε η συνάδελφο δεν ισχύει και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να κινηθούν στο ίδιο μήκο κύματο. Και αν δεν υπάρχει περιθώριο για συμβασμό, τότε θα με όλου του κοιόδε, ώστε να δούμε ποιε θα είναι οι κόκκινε γραμμέ μα. Κατά τα άλλα θα εγκριθεί το σχέδιο κειμένου για πρώτη ανάγνωση, θα ακολουθηθεί η διαδικασία και αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε προ του τέλους της τρέχουσης θητείας. Ελπίζω όσο θα υπάρξει περιθώριο για να μπορέσουμε να συμβαστούμε με το Συμβούλιο και να αντικαταστήσουμε έτσι την ε, απόφασή του. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κοέγιο. Ερχόμαστε λοιπόν εσύ στο σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη. Να διακόψουμε λίγα λεπτά γιατί δεν βλέπω την εισηγήτρια. Έρχονται, έρχεται. Υποτίθεται ότι αρχίζει στις 12 το θέμα αυτό. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 5-6 λεπτά και να αρχίσουμε και πάλι στις 12. Colleagues, I, I propose that we resume. Να ξαναρχίσουμε, συνάδελφοι, σας προτείνω. Λέει πρόεδρος. Okay, colleagues, we continue with point 11 on the agenda. Listing the third countries whose national... Για να δούμε τώρα εδώ το επόμενο θέμα το οποίο είναι η κατάλληλο αυτών των ε, τρίτων χωρών ε, σε σχέση με τι θεωρίε διαβατήρων πρέπει να έχουν ε, οι ηθαγενεί υπήκοοι αυτών των χωρών όταν διασχίσουν τα σύνορα των κρατών μελών και ποιοι εξαιρούνται αυτέ τι ρυθμίσει. Έχουμε εδώ πέρα τώρα κάποιε τροπολογίε οι οποίε έχουν υποβληθεί και η συγγήτρια είναι η κυρία Γκάμπριελ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Σα δίνουμε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Ευχαριστώ τους και ηγητές, την Προεδρία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον επικοδομητικό διάλογο το μένει είχαμε από τότε που ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, ούτω ώστε τώρα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με, με μεταλόγου γνώσεω. Και επίσης ε, θα πρέπει να ευχαριστήσω και του συναδέλφου, οι οποίοι κατέθεσαν τι τροπολογίε του, διότι ε, η αφετηρία μα σήμερα είναι η συζήτηση που έγινε στη Λίμπε. Η πρώτη συζήτηση, οπότε και σήμερα πρόκειται να επικεντρωθούμε ε, μόνο στι ε, τροπολογίε σα. Ε, επίση, ότι ευθύ εξ αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα πρότεινε να διαγράψουμε την υποχρέωση των θεωρήσεων διαβατηρίων για, του 16 χώρε από Καραϊβική και Ειρηνικό και επίση για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία Βρετανών υπηκών. Οπότε έχουμε αυτή τη ρύθμιση σε αυτό το σχέδιο έκθεσης και ε, έχουμε την ίδια λίστα και και σε σχέση με κάποιους ε, Ινδούς όσον αφορά την εξαίρεση από τις φυλές διαβατηρίων. Οπότε έχουμε τώρα 16 τροπολογίες, 8 τροπολογίες οι οποίες έχουν ε, κατατεθεί. Ε, Εμμυράτα ε, επίσης έχουμε το κείμενο 739 του 2001 και υπενθυμίζω ότι η Ιρλανδική Προεδρία είχε θέσει πρώτα το, ε, θέμα τον Ιανουάριο σαν τα μοίρα της διαπραγματεύσεις όσον αφορά τον διάλογο ο οποίος ξεκίνησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οπότε και ήρθαν σε επαφή και με την συγκεντριά σας από τον Μάιο οπότε και έτσι είχαμε σε τακτά διαστήματα επαφές και μπορέσαμε να αποσπάσουμε περισσότερες πληροφορίες περισσότερες λεπτομέρειες οπότε και κατά αυτόν τον τρόπο ε, συνειδητοποίησαμε ότι οι εκπρόσωποι των Εμμυράτων επανειλημμένα ε, είπαν ότι θα ήθελαν έτσι να συσφίξουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Euh, Πέραν όλων αυτών, τώρα θα πρέπει να σας πενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβουλίο είναι οι συνομοθέτες εν προκειμένου από αυτό το οποίο χρειάζεται είναι από κοινού να προβούν τις διαπραγματεύσεις για αυτόν τον, την ανθεώρηση του κανονισμού όσον αφορά την χαλάρωση του κανονισμού για τις θεωρήσεις. Τώρα για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις τροπολογίες. Είναι οκτώ από πλευράς τεχνικής Τέσσερις τροπολογίες χρειάζονται για να φύγει μια χώρα από την αρνητική λίστα στην, στην, στην θετική και έχουμε δύο ομάδες ε, βουλευτών 63 ε, συνολικά που θέλουν να καταργηθεί η θεωρία για τους υπηκόστων των, ε, α, των, των Εμμυράτων και έχουν ε, κατεβάσει τις τροπολογίες. Ναι, έχουμε επομένω σε αυτές τις πληροφορίες και ήρθα σε επαφή με την αυτοεξοχότητα των, των πρέσβη της χώρας και έχουμε αυτό το έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει φόβος λαθροντάφησης, γιατί έχουμε ένα εκατομμύριο αυτών οι οποίοι καλύπτονται από αυτήν την, ε, την απελευθέρωση της βίδας. οπότε γίνεται, γίνεται αυτή η κίνηση και αυτά τα ταξίδια για τουρισμό, για εμπόριο, για οικονομικές σχέσεις με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, οπότε και γι' αυτό και θέλουν να γίνει αυτή η ρύθμιση. Έχουμε 50 δις ευρώ όσον αφορά ε, τις, τις ανταλλαγές με τις, ε, μεταξύ νομιζόντων και χώρες. Έχουμε 160.000 ε, Ευρωπαίους από την Ένωση που μένουν εκεί πέρα. Το, το 2012 είχαμε ένα εκατομμύριο 600.000 περίπου επισκέπτες Ευρωπαίους ή στα Εμμυράτα. Από την άλλη μεριά ε, έχουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση, αλλά έχουμε άλλα δύο θέματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Αφενός θα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη, την ισορροπία, την περιφερειακή που είναι πάρα πολύ βασική. Και θέλουν τα μοιράτα επομένω για να υπάρχει ισορροπία ό,τι, ε, ό,τι πρόβλημα έχει το Ισραήλ. Και επίση είναι και το θέμα τη αμοιβιότητα. Να το δούμε καλύτερα. Ο πρέσβη μου είπε ότι τα Εμμυράτα προθυμοποιούνται να προσχωρήσουν αυτή την αμοιβαιότητα εάν εμείς κάνουμε αυτή τη ρύθμιση για τα Εμμυράτα. Και όταν μιλάμε για 100% αμοιβαιότητα, προκύπτει ότι σήμερα έχουμε δύο διαδικασίες για χορήγηση θεωρήσεων που τα Εμμυράτα εφαρμόζουν όσον αφορά τους Ευρωπαίους. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια προστευμένη διαδικασία ε, που γίνεται δωρεάν για 30 χώρες, μεταξύ των οποίων παλές 15 χώρες μέλη. Σε αυτή την ομάδα έχουμε επίσης και κάποιες χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι στο Σέγγεν. Νορβηγία, Αλβετία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν. Επίσης έχουμε και κάποιες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μονακό, Βατικανό, Σαν Μαρίνο και επίσης χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Επίρου ΕΙΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Μπρουνέη, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Νότια Κορέα, Χονγκ Και πάντως όλες οι άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και τα νέα κρατημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13 δηλαδή ε, έχουν να περάσουν μια πιο περίπλοκη διαδικασία που δεν είναι δωρεάν. Και είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να εξεταστεί καλύτερα, θα πρέπει να δούμε το, πώς θα τηρηθεί η αμοιβαιότητα. πρέπει να τηρηθεί αυτή η αρχή. Αλλά επίσης θα πρέπει να τηρηθεί και η αρχή της μεταχείρισης. Και έχουμε επομένως εδώ δύο κατηγορίες Ευρωπαίων σε σχέση με τη διαδικασία και σε σχέση με το τέλος που καταβάλλει για τη θεώρηση. Ενώ εμείς από πλευράς μας δεν χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες τους υπηκόους των Εμμυράτων. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ε, σπουδαίο πριν ολοκληρωθεί η διεκπαιρέωση του θέματος να θυμιστεί το ζήτημα που σας εξέθεσα. Πάντως, θετικά είναι τα μοιράτα όσον αφορά το να υπάρξει μια κοινή διαδικασία, απλουστευμένη και δωρεάν για όλους τους Ευρωπαίους. Επομένως, θα πρέπει να προσέξουμε αυτή τους την πρόθεση. Και αν συνεχίσουμε την εκπαίδευση του θέματος και γι' αυτό και σήμερα θα ήθελα να ακούσω τι πρεσβεύουν οι άλλες πολιτικές ομάδες. Έτσι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια θέση του Κοινοβουλίου, γνωρίζοντα τα πράγματα ακριβώς όπως γίνεται για όλα τα θέματα. Τα πιο δύσκολα, τα πιο λεπτά. Γιατί όλοι εδώ οι εμπλεκόμενοι διακυβεύουν πολλά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και περιμένω τα σχολεία σας. Ευχαριστώ κυρία Γαβριέλ. Η κυρία Φαγιόν είναι η πρώτη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τη συνάδελφο την κυρία Καπρίελ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Επίσης ευχαριστώ και τους υπολείπους και όδες ε, αυτού του θέματος. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ λίγο στις τροπολογίες που αναφέραμε. Το θέμα των ε, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θα ήθελα να ε, αρθεί η υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίων και να διευκολύνεται ε, η μετακίνηση των ανθρώπων. Αυτό αφορά και επιχειρηματίες και τον απλό κόσμο. Δεν ξέρω αν ε, έπρεπε να περιμένουμε τόσο καιρό, δεν ξέραμε υπήρχε κάποια ρευσότητα στην περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δεν ξέραμε αν θα θέλανε να ενταχθούν τα Εμμυράτα. Ε, ανατράπηκε λίγο η κατάσταση, αλλά τώρα υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια, τη συμπερίληψη δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο θετικό κατάλογο. Πέρυσι Όταν ρωτήσαμε τα κράτη-μέλη αν συμφωνούν να μπουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, απάντησαν μόνο τρία. Τα υπόλοιπα ήταν σε λίθαργο. Μόνο τρία κράτη απάντησαν καταφατικά για συμπερίληψη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο θετικό κατάλογο. Δεν, ναι, έχει νόημα τώρα να χάσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να δώσει το πράσινο φως στη συμπεριλήψη των ΗΠΑ σε περίπτωση που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνήσουν. Πολλοί συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες έχουν πολύ θετική άποψη. Τώρα να δούμε και τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η συμφωνία. Γενικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πληρούν τα περισσότερα κλητήρια. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί σε αυτό. Για να είμαι ειλικρινή, θα πρέπει να πω ότι προς το δικό μα συμφέρον είναι να συμπεριλάβουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι σημαντικό εταίρο μας, στέλνουν πολλούς τουρίστες και δεν συνιστούν οι υπήκοοι τους ε, απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε είναι ελαφρομετανάστες. Υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα. Θα ήταν η μόνη αραβική χώρα που θα συμπεριλαμβανόταν στο θετικό κατάλογο σε χώρες που δεν χρειάζονται οι πολίτες τους θεώρηση διαβατηρίων. Η μόνη μου επιφύλαξη, αν θέλετε, εδώ είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν είμαι η μόνη που έχω επιφύλαξει από αυτού. Αν συγκρίνουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με άλλες χώρες, Μαλαισία επί παραδείγματι, η κατάσταση είναι καλύτερη εκεί. Είχαμε επαφές με τους ηθινόντες μας είπαν τι έχουν κάνει μέχρι τώρα οι κάθε είχε μέχρι και το προνόμιο να εγκαινιάσει ε, το διάλογο για το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, δέχτηκε όλες τις διαβεβαιώσεις ε, από πλευράς των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι ο διάλογος αυτός θα υποστηριχθεί πλήρως και από εκείνους. Η κυρία Γκαμπριέλ μίλησε για την αρχή της αμοιβαιότητας Η αρχή της αμοιβαιότητας τι είναι. Είναι κάτι που υποστηρίζουν και άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι πλέον έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ε, θέμα είναι τώρα να υποστηρίξουμε τις ε, τροπολογίες, θα το συζητήσουμε και στην πολιτική μου ομάδα. Ευχαριστώ κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πάρω το λόγο στη θέση του Μισελ, ο οποίος είναι ο σκιώδης για τους φιλελευθέρους και ο οποίος είναι στη Ρουάντα αυτή την εποχή. Θα σας διαβάσω λοιπόν την παρέμβασή του. Γνωρίζουν οι υπόλοιποι σκιώδης ε, την ε, θέση του βέβαια για τις τροπολογίες. Σχετικά τώρα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει καμία παρατήρηση και καμία αντίρρηση. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ υποστήριξε τις προτάσεις της Επιτροπής όπως και γενικότερα η ομάδα. Μετά από την τελευταία συζήτηση στην Επιτροπή υπήρξαν ορισμένες τροπολογίες στον λεγόμενο θετικό κατάλογο λέγει ότι θα συμφωνήσω με τα προτινόμενα θέματα. Πρώτον ότι τα Εμμυράτα δεν παρουσιάζουν προβλήματα σχετικά με, τους, με την παράνομη μετανάστευση και την ασφάλεια. Έχουν μακρόχρονες σχέσεις με πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, θα πρέπει να διαβηθούν οι σχέσεις αυτές. Τρίτον, χορηγούν βιομετρικά διαβατήρια στους πολίτες τους και θα προσφέρουν μια πλήρη, ε, θα έλεγα, αμοιβαιότητα στις χώρες της Ένωσης. Για τα Εμμυράτα η άρση της α, θεώρησης θα διευκολύνει τις εμπορικές σχέσεις και τις ανταλλαγές της φοιτητικέ. Αυτές είναι οι θέσεις του συναδέλφου. Προσθέτει όμως ότι η ομάδα Δημοκρατών και Φιλελευθέρων δεν έχει πλήρως ακόμα πάρει την τελική της θέση και περιμένει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής. Ευχαριστώ κύριε Γκρίσμπεκ. Τελευταίο αίτημα. Thank you, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι από τους συντάκτες των τροπολογιών. Ε, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια ε, για το έργο της. Έχει ήδη εξηγήσει ε, όλες τις ε, πιθανές ευεργετικές συνέπειες. Ξέρετε ποιοι είναι εκείνοι που επισκέπτονται τα Αραβικά Εμμυράτα ή και ποιοι έρχονται από τα Εμμυράτα στην Ευρώπη. Έχουμε εκπαιδευτικέ ανταλλαγέ ε, και είναι σημαντικό για μα και ακαδημαϊκές ανταλλαγέ για να έχουμε και περισσότερη επιρροή μεθαύριο στα Εμμυράτα. Αλλά έχουμε και εμπορικέ σχέσει που συσφίγονται όλο και περισσότερο ε, με τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι πολύ σημαντικό επίση και θα είναι και η πρώτη αραβική χώρα ε, που θα δει να έρεται υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου και επίσης πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αραβικό κόσμο και είναι και γεωστρατηγική σημασία σε αυτός ο γεωγραφικός χώρος. Καλό είναι λοιπόν να αυξηθεί η επιρροή μας εκεί. Εγώ είχα συζητήσεις με εκπροσώπους ε, της ε, πρεσβείας και του προξενείου στη Βαρκελόνη και είναι έτοιμοι να δεχθούν ε, αυτό με πλήρη αμοιβαιότητα για τις θεωρήσεις και νομίζω αυτό είναι ο τρόπος που θα πρέπει να προχωρούμε και να λύνουμε αυτά τα προβλήματα της διτής εκπροσώπησης ε, με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και με αυτή την εξαίρεση λύνεται. Υποστηρίζω απολύτως λοιπόν την τροπολογία που έχει κάνει ο συνάδελφος Μάριο Ντάβιντ και πολλά άλλα μέλη έχουν συνυπογράψει και νομίζω ότι μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ η Πρόεδρος. Ε, θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία αν θέλουν να ε, σχολιάσουν και μετά η εισηγήτρια να κλείσει και ελπίζω να προλάβουμε μέχρι το 12.30 να τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Το αργότερο. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, έχει το λόγο εκπρόσωπος. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχει περάσει η ώρα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και πάλι ε, για τη θετική της ε, έκθεση και για την τοποθέτησή της. Καλωσορίζουμε πάρα πολύ τη θετική στάση της εισηγήτριας, το είπε και η κυρία Φαγιόν και το ε, θύμισε, η πρόταση για συμπερίληψη των Εμμυράτων στη θετική λίστα είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι το οποίο μπορεί να υποστηρίξει βεβαίω με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει και το Συμβούλιο στην προσθήκη αυτή. Για τα Εμμυράτα νομίζω συμφωνούμε όλοι, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένω σύντομα να αναφερθούμε στο θέμα αυτό της αμοιβαιότητας. Η συγγήτρια ανέφερε κάτι ε, για ελεύθερη κοινοτική διαδικασία. Τι θα πει αυτό ακριβώς. Για την άρση θεώρησης, τη διμερή, αυτή τη θέση ισχύει μόνο εφόσον συναυτεί συμφωνία διμερής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εμμυράτων. Βεβαίως με πλήρη αμοιβαιότητα από τη στιγμή εκείνη ε, και μετά. Τι σημαίνει αυτό. οποιαδήποτε διαδικασία μετά ε, ε, καταργείται γιατί αντικαθίσταται από το νέο σύστημα. Το κατανοούν πολύ καλά και τα Εμμυράτα αυτό και ήθελα να το θυμίσω. Το καταλαβαίνουν και τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσιλωμένη σε αυτή την κατεύθυνση. Και η αμοιβαιότητα μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω μόνο. Ε, προσβλέπω στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέστε. Ευχαριστώ εξ ονόματος της Προεδρίας. Ο κύριος Γιάκη Μαβίτσιος, παρακαλώ. Thank you, Madam Chair, and, and on behalf of the President, also many thanks for the rapporteur for, for, for, for the report. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση και σας τονίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για το Συμβούλιο. Άλλων υπόψη όλες τις τροπολογίες και πρέπει να σας πω ότι όλα είναι και περισσότερα κρατημέλη ε, προστίθεται στους καταλογίνων που θα εγκρίνουν το κείμενο. Πότε περιμένουμε πώς και πώς το τελικό σας κείμενο και ελπίζω ότι σύντομα θα τα βρούμε. Ευχαριστώ και πάλι κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο να πω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που εξέφρασαν τη θέση τους. Επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διευκρινήσεις ε, ε, για το ότι όλα αυτά θα τεθούν σε ισχύ μετά την υπογραφή της Διμερούς Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμμυράτων. Ε, ευχαριστώ την Προεδρία και εκ των προτέρων ε, που μας στηρεί ενήμερους και θα παρακαλώ να μας στηρεί εγκαίρως ενήμερους για την πρόοδο των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλοι έχουμε καταλάβει ότι θα πρέπει να προχωρούμε σε αυτό το θέμα με τα λόγου γνώσεως, να έχουμε συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες κάθε φορά ε, το ξέρουν αυτό και η Πρεσβεία και τα Εμμυράτα. Ε, θα πρέπει να συνεχίσουν να μας ενημερώνουν. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Πάντα γνωρίζοντας ότι η πλήρης αμοιβαιότης και η εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εμμυράτων είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα πρέπει να τηρείται. Και είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη και με αυτό το θέμα. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε να έχουμε μια θέση που θα μας επιτρέψει να αποφαθούμε γνωρίζοντας την κατάσταση και στέλνοντας ένα μήνυμα ισχυρό και ηχηρό, πολιτικό, οικονομικό και κυρίως προς την κατεύθυνση των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει σε μια ημερομηνία που ακόμα απομένει να καθοριστεί. Ε, ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίασή μας. Να ξανάρθει όμως το απόγευμα στις 3 η ώρα παρακαλώ, γιατί έχουμε ακρόαση για τη μαζική ε, παρακολούθηση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας. Επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ.